Okej, okay, eh, Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Να σας καλωσορίσω όλους θερμά στην ε, πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για φέτος. Ως συνήθως, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα και αύριο. Το πρώτο θέμα ήταν η συνεδρίαση των ε, συντονιστών, η οποία ήδη έχει πραγματοποιηθεί και κλεισμένων των θυρών. Το σημείο 2. Σας παρακαλώ, μπορείτε παρακαλώ να καθίσετε. Το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για τροποποίηση. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Προχωράμε στο σημείο 3. Ανακοινώσεις του Προέδρου. να σας ανακοινώσω. Καταρχήν ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές προσωπικού στην ε, Επιτροπή μας μέσα σε δύο μήνες. Θα χάσουμε δύο από τα, από τα μέλη του προσωπικού μας. Η κυρία Σλέντακ δεν θα είναι μαζί μας στην επόμενη συνεδρίαση. Λυπάμαι πάρα πολύ που μας εγκαταλείξεις. Ε, εκτιμούμε πολύ τις ικανότητές σου. Λίγο χαίρομαι που θα παραμείνεις τουλάχιστον στο κοινοβούλιο. Ε, θα εργάζεσαι για την Επιτροπή Πολιτισμού από εδώ και μπρος. Ε, και ελπίζω ότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Πολιτισμού πάνω σε θέματα ισότητας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θητεία σου εδώ και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην καινούργια σου θέση. Επίσης, θα καλωσορίσουμε δύο νέα πρόσωπα. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την κυρία Ταμπορίνη που βρίσκεται Καλά, ας καλωσορίσω πρώτα την κυρία Κόντε Περέιρα. Ορίστε η κυρία Ταβουρίνη, νέο μέλος του προσωπικού. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και καλωσορίζω και την κυρία Κόντε Περέιρα. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας. Λυπόμαστε που χάνουμε ικανούς συνεργάτες, ε, χαιρόμαστε όμως ε, ότι έρχονται νέοι συνεργάτες ε, που θα πάρουν τη θέση τους. Το άλλο θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι ότι θα γίνει τροποποίηση στη... στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής μας λόγω του ότι το Κοινοβούλιο Ε, θα έχει δύο ολομέλειες τον Οκτώβριο. Ε, ε, θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Θα έχουμε πάντως νέες ημερομηνίε για τον Οκτώβριο. Πάντως την Άνοιξη δεν αλλάζει τίποτα. Σημείο 4 στην ημερησία διάταξη. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Έχετε τα πρακτικά της 17ης ε, ε, Δεκεμβρίου. Ε, εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Ωραία. Προχωράμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, που είναι το πρώτο θέμα επί της ουσίας. Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα της γυναίκας. Είναι ένα θέμα που επέλεξε και η Επιτροπή μας ε, για ε, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας που γιορτάσαμε στις 7 Μαρτίου, όχι στις 8 Μαρτίου. Ε, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα την έκθεση αυτή. Η είναι η κυρία Ελίσσα Μωρίν Σαρτιέ. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες, τις οποίες θα συζητήσουμε τώρα. Με πολύ χαρά, λοιπόν... Δίνω το λόγο στην Αντιπρόεδρο, την κυρία Μωρίν Σαρτιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ παρόντες και παρούσες για να ακούσετε αυτή την έκθεση η οποία μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εάν λάβουμε υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι και αν λάβουμε υπόψη επίσης το γεγονός ότι δεν βλέπουμε στο άμεσο μέλλον έξοδο από την κρίση. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική διότι παρουσιάζει τον αντίκτυπο της κρίσης στις γυναίκες και με αυτόν τον τρόπο απεικονίζει ε, την ουσία της εργασίας των γυναικών σήμερα και μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι η φτώχεια είναι γένους θηλυκού και ότι οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη έχουν ακόμα πιο αρνητικό αποτέλεσμα και επίπτωση στις γυναίκες, ε, στις προσωρινές συμβάσεις, στις συμβάσεις μερικής εργασίας, σε όλες δηλαδή τις μορφές εργασίας οι οποίες είναι και οι πιο επίφοβες και οι πιο πρόσκαιρες ε, κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης. Γνωρίζετε ότι στην προσπάθεια αυτή επανένταξης στον χώρο της απασχόλησης πολλών οι οποίοι έχουν τεθεί στο περιθώριο λόγω της κρίσης και άρα πολλών και γυναικών, η πολιτική διαβίου εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και ικανοτήτων, όλα αυτά αποτελούν ένα κινητήριο μοχλό ώστε οι γυναίκες να ανέβουν επίπεδο. Η έκθεση μας δείχνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ως προς τη χρήση αυτού του κινητήριου μοχλού, τον οποίο πιο εύκολα χειρίζονται οι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες, δεδομένου του μεγάλου φόρτου εργασίας των γυναικών. Κατά τρίτο λόγο, η κρίση δείχνει ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε μια πρώτη θέση απασχόλησης, στην πρώτη τους δουλειά. Δυσκολεύονται επίσης να έχουν πρόσβαση στη θέση λήψης αποφάσεων. Δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση ε, στο επιχειρήν, με την ευρεία έννοια του όρου αυτού. Για τον λόγο αυτό, η έκθεσή μας καταλήγει σε διάφορες συστάσεις όσον αφορά σε πολλούς και διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, πράσινη οικονομία, κοινωνική οικονομία, πολιτική μεταφορών. Πρέπει όλες οι προσπάθειες σε όλους αυτούς τους τομείς να συγκλίνουν έτσι ώστε να απαλυνθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης της γυναίκες. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό ήθελα να πω και είναι το εξής. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε είδους πολιτική η οποία θα μας βοηθήσει να συμφιλιώσουμε την προσωπική οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Ιστερούμε πολύ από το να υλοποιηθούν ε, οι προσδοκίες μας. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές συμφιλίωσεις οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν αδύρυτη ανάγκη και κατά τη διάρκεια ε, της ανατροφής των παιδιών στην πολύ μικρή τους ηλικία αλλά και κατά τη διάρκεια φροντίδας των ηλικιωμένων διότι πολύ συχνά και για λόγους πολιτιστικούς αν θέλετε η γυναίκα σε μια οικογένεια επιβαρύνεται περισσότερο με όλα αυτά τα βάρη και έτσι απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το χώρο εργασίας. Οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη σήμερα δεν λαμβάνουν τόσο υπόψη τους τη δυνατότητα πλαισίωσης των παιδιών σε πολύ μικρή και νεαρή νηπιακή ηλικία, μικρότερη της νηπιακής ηλικίας και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να υποδεχθούν παιδιά κάτω των τριών ετών. Και τέλος θα ήθελα να επιμείνω σε αυτές τις προκαταρκτικές σκέψεις που σας παρουσιάζω στην απουσία ενός ε, οδικού χάρτη αν θέλετε, απουσία παρατήρησης παρακολούθησης του τι γίνεται με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αναφύλο ε, τις εξελίξεις, τον αντίκτυπο στους άνδρες και στις γυναίκες, τον αντίκτυπο που έχει κρίση και πώς εξελίσσεται αυτή ε, και πώς εξελίσσονται και αλλάζουν οι επιπτώσεις και στους άνδρες και στις γυναίκες. Και ε, νομίζω ότι αυτό θα μας αποκάλυπτε πολλά αποκαλύπτει καταρχάς την απουσία βούλησης επίλυσης όλων αυτών των προβλημάτων υπό το οπτικό πρίσμα της πλήρους ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, στον χώρο εργασίας γενικότερα. Στην έκθεση λοιπόν που σας παρουσιάζω, ε, μετά τη γνωμοδότηση και της κυρίας Τζίμερ από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση άλλωστε με τη δική μας, και νομίζω ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ε, το ότι δηλαδή η Επιτροπή για τις Γυναίκες και την Ισότητα των Φίλων και η Επιτροπή για την Απασχόληση ε, υιοθετούν απόψεις οι οποίες συγκλίνουν απολύτως ως προς τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. 279 τροπολογίες, 70 από τους σοσιαλιστές, 63 από το ΕΛΚ, αλλά και εγώ ίδια προσωπικώς υπέβαλα τροπολογίες στο δικό μου σχέδιο ε, ε, έκθεσης, 24 από την 24 τροπολογίες της ΓΚΟΕ, ο κύριος Πρόεδρος Κούσταυσον της Επιτροπής μας ε, έκανε πολλή δουλειά, προσπάθησε πάρα πολύ να υποβάλει τροπολογίες στην έκθεση αυτή και τον ευχαριστώ. 15 τροπολογίες από την Άλντε, 4 από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και 3 από τους πράσινους τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους για τις τροπολογίες αυτές. Βλέπω και ερμηνεύω την υποβολή τροπολογιών ως έκφραση και εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευρά σας ε, για ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους και που σίγουρα μας απασχολεί όλους. Πιστεύω σε γενικές γραμμές ότι όλοι επιθυμούμε οι γυναίκες να ενταχθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας και οι θέσεις απασχόλησής τους να είναι όσο πιο σταθερές γίνεται. Ανεξαρτήτως ε, του πού τοποθετούμεθα στο πολιτικό φάσμα ή μεν ή δε, αυτό που σίγουρα μας ενώνει, το κοινό στοιχείο μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και το κοινό στοιχείο μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν υποβάλει τροπολογίες είναι ακριβώς αυτό, η βούλησή τους οι γυναίκες να ενταχθούν με σταθερό και βιώσιμο τρόπο στην αγορά εργασίας. Εάν έχουμε αυτό ως αφετηρία, σίγουρα θα μπορέσουμε να χαράξουμε συγκλίνουσες και όχι αποκλίνουσες γραμμές. Επομένως, ε, η έκθεση αφορά στην πρόσβαση στην εργασία, αφορά στη σταθεροποίηση των συμβάσεων εργασίας, τη μονιμοποίηση δηλαδή, την καταπολέμηση της μη αμοιβόμενης εργασίας, την ισότητα ε, των μισθών, την εξάλληψη των μισθολογικών ανισοτήτων και την εξάλληψη των ανισοτήτων ως προς την εξέλιξη, την επαγγελματική και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι βασικοί άξονες και όλες οι τροπολογίες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να υπάρξουν συμβιβαστικέ λύσεις. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο άλλωστε συγκροτεί και την κοινή άποψη, το κοινό όραμα που έχουμε όλοι για το θέμα αυτό, είναι το εξής Έχουμε βούληση, τη βούληση να κάνουμε το παν η εργασία να χειραφετεί τις γυναίκες, να τις καθιστά αυτόνομες. Και πρέπει να το υπενθυμίσουμε, διότι αυτό είναι και ο πολιτικός στόχος. Στην ισότητα των πολιτών θα πρέπει οι γυναίκες να είναι αυτόνομες, επί ίσης με τους άλλους πολίτες, μέσω της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι το σύνολο των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί σε αυτό το σχέδιο έκθεσης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και από τις τροπολογίες αυτές ε, καταλήγω σε ένα δεύτερο σημείο το οποίο ε, θα μας σε αυτό το δεύτερο σημείο το οποίο θα μας κάνει πραγματικά να βρούμε ένα κοινό τόπο μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων. Τρίτη παρατηρήση, ο αντίκτυπος των πολιτικών λιτότητας. Το θέμα αυτό μπορεί να διατυπωθεί με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι σίγουρο μπορούμε να το διατυπώσουμε υιοθετώντα ε, πολύ με έντονα πολιτικό λεξιλόγιο ή πολύ έντονα οικονομικό λεξιλόγιο ή πολύ έντονα κοινωνικό λεξιλόγιο. Όπως και το διατυπώσουμε όμως, ε, δεν υπάρχει απόκληση στη συμφωνία μας, πιστεύω. Ίσως, κύριε Πρόεδρε, θα σας άρεσε εσάς να έχουμε αποκλίνουσες απόψεις για το θέμα αυτό. Όμως είναι πασιφανές ότι σε όλους είναι υποσύφανε ότι οι πολιτικές λιτότητες ε, αποτέλεσαν απαραίτητο και σημαντικό παράγοντα μέσω του οποίου αυθορμήτως οι γυναίκες ε, τέθηκαν στο περιθώριο. Ορισμένες γυναίκες αυθόρμητα αποσύρθηκαν από το χώρο εργασίας δεν λέω ότι παντού συνέβη αυτό, αλλά η κρίση οδήγησε στο να τεθούν τόσο στο περιθώριο από την αγορά εργασίας πάρα πολλές γυναίκες, είτε λόγω των εξελίξεων, είτε τελικά μέχρι και ε, αυθορμήτως. Σε μία πρώτη φάση δεν επλήγησαν οι κλάδοι της οικονομίας όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, ωστόσο οι πολιτικές λιτότητες των κρατών πλήττουν ιδιαίτερο τους κλάδους της ε, οικονομίας όπου κυριαρχούν οι γυναίκες σε δεύτερο χρόνο. Και αν προσθέσουμε κιόλας και τις γυναίκες που οι ίδιες αποσύρονται λόγω της κρίσης από την αγορά εργασίας, βλέπουμε τον τεράστιο αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας ε, στις γυναίκες. Όπως και να το διατυπώσουμε λοιπόν, ε, με δογματικό τρόπο, με πολιτικό, με κοινωνικό ή με οικονομικό τρόπο, όποιες λέξεις και αν βρούμε, πάντοτε ε, το ίδιο μήνυμα είναι αυτό που εκπέμπουμε, ότι δηλαδή οι πολιτικές λιτότητες έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο ε, στην κατάσταση των γυναικών σήμερα. Τέταρτο σημείο που πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση είναι το εξής. Η διαφοροποίηση εντός Ευρώπης, εντός ε, χωρών μελών μεταξύ π.χ. των γυναικών από το βορρά και των γυναικών από το νότο. Η Αντιγόνη έχει υποβάλει για παράδειγμα μια τροπολογία ε, προς αυτή την κατεύθυνση και άλλοι επίσης και άλλες. Βλέπουμε λοιπόν ότι διευκρινίζεται ιδιαιτέρως η κατάσταση των γυναικών στο Νότο, στο σχέδιο έκθεσής μας. Και αυτό είναι κάτι που με άγγιξε προσωπικά και ε, δεν είναι δυνατόν να μην το λάβω υπόψη μου. Προφανώς. Τώρα, πολλές τροπολογίες, αρκετές μάλλον, έχουν να κάνουν με αυτό που ανέφερα πρώτο. Η ισότητα μεταξύ πολιτών ε, οδηγεί στο να είναι αδύρυτο το δικαίωμα ε, των γυναικών στην εργασία. είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμμερίζονται όλες οι χώρες της Ευρώπης και η δική μας δουλειά θα πρέπει να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός, ώστε πράγματι να οδηγηθούμε ως κοινωνίες σε αυτή την ισότητα, την πλήρη μεταξύ πολιτών, όπου όλοι θα έχουν ακριβώς το ίδιο δικαίωμα στην εργασία. Τώρα, ως προς τις γυναίκες και τη σταδιοδρομία. Έχοντας τη βούληση να προβάλλουμε την ανάγκη για την μισθολογική ισότητα αλλά και για την ίση, ίση πρόσβαση στην επαγγελματική εξέλιξη και ανέλυξη στη σταδιοδρομία, ορισμένοι εξημών με υψηλών έχετε υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και στις τροπολογίες προβλέπετε πιο συγκεκριμένα ότι οι γυναίκες δεν είναι ενταγμένες, δηλαδή είναι αποκλεισμένες, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις θέσεις όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και κυρίως όχι σε όλους τους κλάδους ε, της οικονομίας. Σε καιρούς λοιπόν οικονομικής κρίσης, κάτω τους οποίους οι αποφάσεις που θα ληφθούν είναι αυτές που θα αναδομήσουν το σύστημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι αποκλείονται οι γυναίκες γιατί δεν είναι παρούσες σε αυτό το σύστημα λήψης αποφάσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, το έχουν ε, τονίσει ε, οι παρεμβαίνοντες στις διάφορες τροπολογίες τους και νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις που θα κινούνται όμως γύρω από αυτό την ε, συμπερασματική παρατήρηση, γιατί ε, θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα πάρα πολλές τροπολογίες έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, με τον αυξημένο ε, κίνδυνο απόλυσης, με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και καθεξής. Με όλα αυτά δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόσκαιρη απασχόληση και ασταθεί σε καιρούς κρίσης. Ε, μία τροπολογία είχε να κάνει με πολύ συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες είναι και πολύ πιο ευπαθείς ε, σε καιρούς κρίσης. Όλες αυτές οι τροπολογίες είναι απολύτως κατανοητές και απολύτως αποδεκτές από τη δική μου πλευρά. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό το καμβά ε, θα δουλέψουμε όλοι. Τέλος, θα ήθελα να επιμείνω σε τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να τονίσουμε την ανάγκη οι γυναίκες να φτάσουν σε θέσεις λήψης αποφάσεων, σε διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις, ώστε να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις σημαντικές εξελίξεις. Οφείλω να πω ότι όσο δεν χρησιμοποιούμε ως εργαλεία τις στατιστικές τους καταλόγους, τις λίστες, ε, τα συγκεκριμένα αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία, τότε τόσο δεν θα μπορούμε να απαιτούμε τα δέοντα από τις ηγεσίε. Θα πρέπει να μπορούμε να ε, παρακολουθούμε με λογιστικό τρόπο, με μαθηματικό τρόπο τα πράγματα για να ξέρουμε και γιατί μιλούμε. Τελικά η πολιτική ζωή προτιμά να μην έχει συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Προτιμά να μην τα βλέπει. η να ήταν η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας επιπρόσθετη δυσκολία που θα πρέπει να υπερπηδηθεί σε καιρούς κρίσης. Αυτό φαίνεται να πιστεύει πολύ συχνά ο πολιτικός κόσμος. Αυτό φανταζόμαστε άλλωστε. Το Μάρτιο διεξήχθη μία έρευνα με αντικείμενο το εξή. Σε καιρούς κρίσης είναι προτιμητέο οι άντρες να έχουν προτεραιότητα στην εργασία και το 63% απάντησε καταφατικά. Ναι, οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην αγορά εργασίας σε καιρούς κρίσης. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν εδρεωθεί η υποχρέωση τήρηση στατιστικών δεδομένων και έχουμε Ινστιτούτο και Ίδρυμα σχετικό και πολλοί από σας θέλουν, θέλουν ρητή αναφορά στο, στη στατιστική υπηρεσία, εάν δεν γίνει παραγωγική δουλειά, επικοδομητική, επιστημονική και συγκεκριμένη, τότε δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε την ισότητα στο χώρο εργασίας στην οποία προσβλέπουμε με την έκθεσή μας. Αυτά κύριε Πρόεδρε, εν συντομία ήταν η, τα σχόλιά μου για τις θεματικές ενότητες τροπολογιών και της έκθεσής μου εκτός από ορισμένες προτάσεις κατάργησης συγκεκριμένων διατυπώσεων, ε, τις οποίες πρότειναν ορισμένες πολιτικές ομάδες και για τις οποίες δεν βλέπω να υπάρχει ομοφωνία στην Επιτροπή, κατά τα λοιπά νομίζω ότι θα, θα καταλήξουμε σε μία ε, ισχυρή έκθεση η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Παπαδοπούλου πρώτα. Yes. Thank you. I think it's working now, isn't it? Okay, <laughs> very good θα ήθελα να συγχαρώ ακριβώς τη συγγραφέα για αυτήν την έκθεση η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της γυναίκε. Είναι γεγονός ότι διαβάζοντας τη ένιωσα την ανάγκη να γίνει ειδική αναφορά στις γυναίκες του Ευρωπαϊκού Νότου και μάλιστα στο γεγονός ότι δεν πλήττονται μόνο οι γυναίκες που εργάζονται στο δημόσιο αλλά και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα γιατί μέσα στην έκθεση γίνεται αναφορά πιο πολύ ότι ετεροχρονισμένα είχαμε θύματα γυναίκες από την οικονομική κρίση, ενώ αρχικά η κρίση είχε χτυπήσει πιο πολλοί άντρες και γίνεται αναφορά ότι χτυπήθηκαν κυρίω γυναίκε που εργάζονται στο δημόσιο. Η δική μα εμπειρία από τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου είναι ότι τα πρώτα θύματα στον ιδιωτικό τομέα που χάνουν τι δουλειέ είναι οι γυναίκε. Διότι έχουν κάποιε συλλογικέ συμβάσει, λόγω τη κρίση οι εργοδότε δεν πληρώνουν κανονικού μισθού, μειώνουν αισθητά το, το μισθό και δίνουν την ευχαίρεια, ρωτούν τι γυναίκε, θέλετε να παραμείνετε με μειωμένο ρυθμό και με αύξηση των ωρών εργασία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετέ δεν μπορούν να μείνουν στη δουλειά, γιατί αύξηση του χρόνου εργασία σημαίνει υποδομέ συμφιλίωση οικογενειακών επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και αυτό είναι κάτι πολύ σωστό που έχετε εντοπίσει στην έκθεση, ότι δεν υπάρχουν οι ίδιε υποδομέ σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Εάν πάντα μιλούμε, όταν μιλούμε business as usual και κάνουμε τροπολογίε σε εκθέσει για θέματα γυναικών, αυτό που πρώτη τα λέμε πάντα είναι να μην θυματοποιούνται οι γυναίκε και να υπάρχουν υποδομέ συμφιλίωση οικογενειακών επαγγελματικών υποχρεώσεων. Λόγω του κύκλου αυτού, του φαύλου κύκλου, τη μείωση ακριβώ τη κρατική φροντίδα, των λεφτών που δίνονται μέσα από του προπολογισμού για να στηριχτούν υποδομέ οι γυναίκε όχι μόνο στιγματίζονται, αλλά όταν θα έχουν την επιλογή περισσότερε ώρε εργασία στη δουλειά ή να μείνουν στο σπίτι, θα αναγκαστούν να μείνουν στο σπίτι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναφορά. Και επιση μια άλλη αναφορά που έχω κάνει στι δικέ μου τροπολογίε είναι ότι οι πάντε μιλούν για μια χαμένη γενιά νέων, ανδρών και γυναικών. Πραγματικά με λυπεί αυτή η φράση, γιατί έχουμε και εμεί παιδιά σε αυτέ τι ηλικίε που έχουν πάρει τα πτυχία του, πρώτο, δεύτερο πτυχίο, προσπαθούν να μπουν στην αγορά εργασία. Είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχουν ίσε ευκαιρίε ούτε για του νέου, ούτε για τι νέε. Και το πρόβλημα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώ το αντιμετωπίζουμε. Επομένω, γίνεται μια αναφορά ότι αυτή η χαμένη γενιά ελπίζω να μην κρατήσει μακρόν η οικονομική κρίση και πράγματι να επανακάμψουν οι οικονομίες για να μπορούν να έχουν θέσεις εργασίας διότι διαφορετικά δεν θα μένουν στι χώρε όπου σπούδασαν για να δουλέψουν, αλλά θα αναγκάζουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό και θα υπάρχει διαρροή εγκεφάλων. Ε, συγχαίρω για την ε, έκθεση και ε, έναν τρίτον είναι η αναφορά ότι δεν υπάρχουν ακόμα reliable statistical data. Είναι κάτι που συζητούμε σε ολέ τι εκθέσει. Θα ήταν καλά να έχουμε συγκριτικά στατιστικά δεδομένα Πώ ακριβώ επηρεάζονται οι γυναίκε στον Ευρωπαϊκό Νότο συγκρινόμενε με τι γυναίκε στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη γιατί όταν έχει αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα και κάνει σωστέ διαγνώσει, τότε βρίσκει και τι σωστέ θεραπείες και τελειώνοντα οι πολιτικές λιτότητας που εφάρμοσαν η Τρόικα δεν έφερα λύσει των Ευρωπαϊκών Νότων ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Πορτογαλία και δυστυχώ και η χώρα μου μπαίνει σε μνημόνιο και πολύ ανησυχώ ότι η ίδια καταστροφή που έγινε στι άλλε χώρε θα γίνει και στην οικονομία τη Κύπρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προφανώς να συγχαρώ την συνάδελφο Μωράν Σαρτιέ για την εξαιρετική της έκθεση και γιατί πρόκειται για ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και τον κατάλογο προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πρόταση της Επιτρόπου Ρέντινγκ, έχουμε γκρίνει ένα τέτοιο κατάλογο στο 2015, καλό όμως θα ήταν να θεωρήσουμε κάποιες από τις προτεραιότητες Και να δώσω απλώς δύο παραδείγματα. Ω προ την Ευρώπη του 2020, μεταξύ των στόχων έχουμε μιλήσει για την απασχόληση των γυναικών και την μείωση της φτώχειας. Εδώ γνωρίζουμε το αντίστροφο φαινόμενο και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή μείωση της απασχόλησης των γυναικών και αύξηση της φτώχειας των γυναικών. Εδώ, στην κρίση, θα πρέπει να δούμε και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιφάσεων και παραδόξεων που προκύπτουν. Όπως είπε και η συνάδελφος Παπαδοπούλου. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ευρώπη ως ε, προς τους κοινωνικούς παράγοντες προστασίας λόγου χάρη για όσους κάνουν την ε, εργασία τους. Υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους νέους θα χρειαζόταν ενδεχομένως ενίσχυση της έκκλησης για εναρμόνιση. Να ενδυναμωθεί το σύστημα αποζημίωσης ε, επιδομάτων ενεργείας, ε, απώλειας της απασχόλησης. Οι γυναίκες στην Ιταλία ονομάζεται αυτό Ταμείο Συμμετοχής όταν μια γυναίκα απευθύνεται στο Ταμείο Ενεργείας. Ε, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματικοί κλάδοι λοιπόν όπου υπάρχει μικρότερη προστασία για τις γυναίκες και αυτό πρέπει να το δούμε. Επίσης, Πρέπει να δυναμώσουμε τις σχετικέ ε, τροπολογίες, αλλά εδώ δίνω έμφαση στο εξή, ότι η χρήση ακόμα και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σημαίνει ότι όταν εμεί εγκρίνουμε το νέο πρόγραμμα θα υπάρξει έγκριση του Ταμείου παραλίλω. Οπότε. Έχω δει εγώ τι έχουν κάνει οι θύνοντε τη δική μου κυβέρνηση, στη δική μου περιφέρεια. Έχουν πραγματικά ασχοληθεί πολύ και με την επιχειρηματικότητα των γυναικών και με την κοινωνική πρόνοια για την προστασία των γυναικών και με, το, με την κοινωνική διάστηση που αφορά τι γυναίκε και το mainstreaming. Εδώ Σημαντικό είναι να τονιστεί επίσης η ιδιαίτερη θέση των ε, γυναικών μεταναστιδών που ζουν στις χώρες μας. Η κοινωνική πρόνοια θα πρέπει να να προωθηθεί στα κοινωνικά συστήματα όλη τη Ευρώπη, αλλά να δούμε και τι μικρέ επιχειρήσει, τι μικροπιστώσει που μπορούν να δοθούν σε αυτέ τι γυναίκε για να τι στηρίξουμε και έπειτα για τα δεδομένα, για την αξιοπιστία των δεδομένων. Ε, εκφράζεται μια ευχή στην έκθεση ότι θα μπορούσε το παρατηρητήριο για την ισότητα των φύλων να αρχίσει να μα δίνει σχετικά συστήματα. Υπάρχει όμω στοιχεία, υπάρχει όμως και γύρω στα, υπάρχουν εθνικά στατιστικολογικά συστήματα Τώρα το να απευθυνθούμε μόνο, για το μόνο στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την ισότητα των φύλων για το θέμα αυτό, δεν αρκεί. Θα πρέπει να διαδικτυωθούμε μεταξύ του οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονε για να δούμε πώ θα αποτιμηθεί ο αντίκτυπο ποιοτικό και ποσοτικό. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μια πιο συγκεκριμένη εντολή στο Ίδρυμα. Η κυρία Βέρμα, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που ήδη άκουσα όσον αφορά την πολιτική λιτότητα και τις γυναίκες. Έχουν γίνει θύματα όχι μόνο στο Νότο και στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που ε, ε, είναι θύματα της πολιτικής λιτότητας. Ε, δεν έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό. Θα πρέπει να γίνουν σχετικές μελέτες, ε, αλλά ε, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε του, του κάθε κράτου μέλου, διότι μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων και να γνωρίζουμε πού ακριβώ βρίσκεται το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική και αναλυτική έκθεσή τη. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντάλοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να πω ότι η συγγέντρια μας παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση. Μεταξύ των σχολείων μου, να πω κάτι που θεωρώ σημαντικό, αν και ακούστηκε και προηγουμένως, ότι λόγω της κρίσης πολλοί χάνουν τη δουλειά τους και μάλιστα όλο και περισσότερες γυναίκες. Πολλέ φορέ είναι οι πρώτε που απολύονται και μάλιστα εκείνε που είναι μεγαλύτερη ηλικία. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Μια άλλη σημαντική πτυχή, ιδιαίτερα στι σημερινέ συγκυρίε, είναι η εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι το 50% των ε, αποφύτων πανεπιστημίων είναι γυναίκε. Όμω μόνο το 40% των θέσεων εργασία δίδονται σε γυναίκε. Υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη απόσταση. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει την πολυτέλεια να μην χρησιμοποιεί το 56% του δυναμικού της, δηλαδή τις γυναίκες. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για γυναίκες καθώς και την εκπαίδευσή τους. Ακόμη και να λάβουμε υπόψη και τι ηλικιακέ διαφορέ. Δηλαδή, η προσπάθεια να κατευθύνεται στι μεγαλύτερε ηλικίε και στι νεότερε οι υπόλοιποι. Ώστε να υπάρχει και μια ανταλλαγή σκητάλη. Δεν θέλουμε επίσης να επικρατήσει η παρουσία των γυναικών στην περίπτωση του φαινομένου της φτωχοποίησης όπως έχει Κατά τα άλλα, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και καλή σας τύχη. Ε, Ευχαριστώ. Να πάρω και εγώ τον λόγο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια. Όπως είπα, όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό τον ε, Δεκέμβριο, πιστεύω ότι έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η έκθεση περιλαμβάνει πολλά σημαντικά θέματα και ε, το ότι υπάρχουν 179 τροπολογίες, ακριβώς όπως είπες, οφείλεται ε, στο μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, δεν είναι δείγμα επίκρισης. Πάρα πολλοί λοιπόν θέλησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Εγώ θα ήθελα η έκθεση αυτή να είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη. Και ήθελα βέβαια και όσο καλή και ε, να πιστεύω ότι είναι, θα ήθελα να ε, συμπεριλαμβάνει το εξή. Ε, η περιγραφή της κατάστασης είναι πολύ καλή. Πράγματι αυτά ισχύουν. Ε, αναφέρεις και τις ε, συνέπειες για άντρες και γυναίκες, και αυτό είναι πολύ καλό, σε τρίτον στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ε, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως που μου λείπει εμένα και δεν θα σε εκπλήξει αυτό που λέω, ε, αυτό που μου λείπει είναι το τέταρτο μέρος, το βασικό πρόβλημα, γιατί βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή. Ο λόγος είναι ότι έχουμε μια πολιτική λιτότητα η οποία επιβάλλει μια πολιτική στην κάθε χώρα χωρίς ε, να μπορεί να προσαρμοστεί η πολιτική αυτή στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι τα άλλα τρία μέρη είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν θα μπορούσα να έχω ε, γράψει καλύτερα τα τρία αυτά μέρη, ε, αλλά εγώ θα ήθελα και το τέταρτο αυτό μέρος. Βέβαια είμαι αριστερός εγώ, οπότε δεν θα σε εκπλήξει αυτό που λέω. Αυτό μου λείπει, διότι χωρίς ένα τέτοιο μέρος... Ε, Μπορούμε με να έχουμε κάποια μέτρα όπως ε, αναφέρεις, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα που είναι η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και που η Κομισιόν επιβάλλει στα, στις διάφορες χώρες. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και σίγουρα το έχεις δει αυτό στις τροπολογίες μου, ε, την επικέντρωση ακριβώς σε αυτές τις οικονομικές πτυχές. Και όσον αφορά τα άλλα τρία μέρη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πρόβλημα να συμφωνήσουμε. Θα βρούμε ε, συμβιβαστικές διατυπώσεις, αλλά ίσως ε, να έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά το τέταρτο μέρος. Ε, και... Ναι, μάλλον πρέπει να δεχτούμε ότι δεν συμφωνούμε απόλυτα σε όλα τα πράγματα, αλλά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την έκθεση, διότι είναι πάρα πολύ καλή. Και δίνω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Ταβόνη. Η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Απλώς να επιστήσω την προσοχή σας σε μία μελέτη. Μελέτη που μόλις ε, δημοσιεύσαμε για τον αντίκτυπο της κρίσης ε, στους άνδρες και τις γυναίκες. Τέλος Δεκεμβρίου ε, δημοσιεύτηκε και την αποστήλαμε στη γραμματεία σας στις αρχές Ιανουαρίου. Δείχνει η μελέτη με τα στοιχεία της ότι υπήρξε αντίκτυπος στις αποκλήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην εργασία και στον μισθό και στην φτώχεια και στην ανεργία. Μειώθηκαν οι αποστάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, όμως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό απετέλεσε πρόοδο προς την επιδίωξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, διότι η κάλυψη των αποστάσεων οφείλεται ακριβώς σε ταχύτερη επιδείνωση της ε, εργασιακής κατάστασης των ανδρών. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για περισσότερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν δεν κανείς τους πίνακες, οι διαφορές ε, μισθών, ε, ποσοστών ενεργείας, απασχόλησης δείχνουν ότι οι διαφορές απλώς περιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί τις διαφορές αυτές και χάρη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτά είχα να πω προς στιγμή. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, ε, να δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Μωρέα Σαρτιέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους και τις συναδέλφους που πήραν το λόγο διότι για ένα θέμα τέτοιο θα πρέπει να οι δικές μας σκέψεις και προθέσεις να ενωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί όθηση στην εξέταση του ε, θέματος. Δεν θέλουμε να αποτελέσει αντικείμενο αντιπαραθέσεων το θέμα αυτό είναι ένας στόχος που όλους μας αγγίζει. Δεν θυμάμαι ποια συνάδελφος είπε ότι τα παιδιά μας ε, σπούδασαν, τα εγγόνια μας επίσης, θέλουμε τα κορίτσια, οι γυναίκες να συσσωρεύουν πτυχία και να μην έχουν δουλειά. Διότι αυτή είναι η σημερινή κατάσταση οι νεαρές γυναίκες έχουν περισσότερα πτυχία από ότι οι συνομήλικοι άντρες. Έχουν όμω μεγαλύτερε δυσκολίε να βρουν δουλειά. Μάλιστα με χαμηλότερου μισθού, με επισφαλέστερες συμβάσει και τελικά λιγότερε πιθανότητε να εξελιχθούν επαγγελματικά. Εδώ λοιπόν η κρίση ε, ουσιαστικά επιτείνει τις δυσκολίες Εδώ λοιπόν θα επιμείνω ε, ώστε όλοι να έχουν πια την βούληση να προσπαθήσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση με επενδύσεις στην εκπαίδευση των ε, γυναικών και δημόσια κονδύλια και ιδιωτικά αλλά και οικογένειες που έχουν ξοδέψει σοβαρά ποσά για την εκπαίδευση των κοριτσιών τους. Είμαι λοιπόν ε, πραγματικά πεπισμένη και το λέω χωρίς να βασίζομαι σε στατιστικά στοιχεία απαραίτητο, αλλά είμαι βαθιά πεπισμένη ότι αν θέλουμε να συμμετάσχουν ενεργά οι γυναίκες στον χώρο εργασίας, θα μπορέσουμε να βρούμε και καλύτερες διεξόδους από την κρίση από ότι το αντίστροφο. Δεν μπορούμε να γνωρούμε ένα τέτοιο όγκο ευφυΐας, ε, δυναμικού παραγωγής η εργασία των γυναικών είναι άκρο σημαντική. Να ξεκινήσω από τη δική σας παρατήρηση, Πρόεδρε, για την σημασία των επιπτώσεων της δημοσιονομικής λιτότητας. Τον έφεραν και άλλες συνάδελφοι των αντικτυπών των αποφάσεων της Τρόικα. Βεβαίως, οι αποφάσεις δημοσιονομικής λιτότητας επηρεάζουν ακόμη περισσότερο και πολύ περισσότερο την εργασία των γυναικών από την εργασία γενικώ. Πλήττεται η εργασία των γυναικών. Στις τροπολογίες που αναφέρατε και έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα, όπως η τροπολογία 17, η τροπολογία 23, η τροπολογία 50 για την ανεξαρτησία των γυναικών. Να πω εδώ, Πρόεδρε, ότι εδώ συμπίπτουν απόλυτα οι απόψεις μας. Το ερώτημά μου, και αν έχετε την απάντηση, ευχαριστώ να την δεχτώ, είναι, στη στρατηγική της Λισαβόνας 2000-2010 γινόταν διαρκώς λόγος για ανάπτυξη. Όμως τότε καθόλου δεν επιταχύνθηκε διαδικασία συμπερίληψης των γυναικών στον επαγγελματικό βίο, τον χώρο της εργασίας. Δίνοντας έμφαση λοιπόν στη δημοσιονομική λιτότητα, στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, στην ανάπτυξη σε αντιπαράθεση με τους στόχους της Ευρώπης του 2020, εδώ κάπως διερωτώμε. Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε πιο χειροπιαστά αποτελέσματα επιλέγοντας τη μία οδό από την άλλη. Άρα, τι μας λείπει σήμερα, τι μας λείπει ώστε να φτάσουμε στην πραγματική συμμετοχή των γυναικών, την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας. Όπως ξέρετε στη χώρα μου συζητάτε αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο για την ισότητα σε επίπεδο εκλογικό. Εάν γνωρίζατε τι έχουμε ακούσει στην Γαλλική Βουλή και στη Γερουσία για το ποσοστό γυναικών ε, στο χώρο εργασίας, θα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για κάτι σκανδαλώδες βλέπουμε ότι υπάρχει βαθιά ριζωμένη αντίληψη μη ισότητας, ανισότητας ε, ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει εδώ να υπάρξει αντιπαράθεση αλλά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τον τελικό στόχο. Άνδρες και γυναίκες να συμμετέχουν με ίσο τρόπο στο χώρο εργασίας με σταθερότητα της εργασίας και με προοπτικές επαγγελματικής ανέλυξης. Νομίζω, Πρόεδρε, αυτά είναι ζωτική σημασίας. Βεβαίως, το παρελθόν δεν μπορούμε να το παρνηθούμε. Υπήρξαν αποφάσεις που δεν ήταν αναγκαστικά συνετές, όμως εγώ τώρα με την έκθεση αυτή θα ήθελα να μην συνεχίσουμε να καθυστερούμε να σέρνουμε το βάρος του παρελθόντος σαν μια μπάλα φυλακισμένου στα πόδια μας. Όχι. Να κάνουμε κάτι για τη συμπερίληψη των γυναικών στον χώρο εργασίας. Και ίσως η κρίση να είναι ακριβώς μια ευκαιρία για να ρίξουμε φως ε, στον πολιτικό αυτό στόχο. Στόχο προς τον οποίο πρέπει να οδηγήσουμε όλα τα κράτη. Τίμησα ιδιαιτέρως, το είπα μόλις, τις ε, παρατηρήσεις της κυρίας Νεβεντάλοβα για την ανεργία και την εργασία των γυναικών. Διερωτώ με τώρα εάν η κατανομή της απασχόλησης μπορεί να γίνει όπως την περιγράψατε και να σας πω ποια είναι και η απορία μου θα μπορούσε να φανταστεί κανείς για να, για να συμμετάσχουν στο χώρο εργασίας άνεργοι άντρες ότι θα γίνει μια τέτοια κατανομή της εργασίας για άντρες. Δεν γίνεται για τους άντρες, ενώ για τις γυναίκες μπορεί κανείς να το σκεφτεί. Καταλαβαίνετε, πρέπει και εμείς οι ίδιες να προσέχουμε ιδιαιτέρως, ώστε να μην προτείνουμε λύσεις που διαφέρουν για την περίπτωση των γυναικών από ό,τι για την περίπτωση των ανδρών. Και κατά κάποιο τρόπο κάνουν ακόμη πιο ευάλωτε στι γυναίκε στο χώρο εργασία. Για την ε, συμμετοχή των πτυχιούχων, ναι, βεβαίω. Ε, πρέπει κάτι να γίνει για αυτέ τι γυναίκε, αλλά τώρα για την κατανομή τη εργασία γυναικών. Γιατί πραγματικά δεν ζητάμε το ίδιο από όλου. Αυτό διερωτώ θα προτιμούσα λοιπόν να υπάρχει αυτή η συμμετοχή, η συμπερίληψη με τρόπο, με γνώμονα την ισότητα. Θα μπορούσαμε όμως να το ξανασυζητήσουμε για να συντονίσουμε τις απόψεις μας. Άκουσα με προσοχή όσο είπε η κυρία Κώστα και η κυρία Παπαδοπούλου για τα προβλήματα των στατιστικών στοιχείων. Καταλήγω και εγώ στο ίδιο συμπέρασμα με σας. Ναι, μα λείπουν τέτοια στοιχεία. Όμω δεν μπορούμε να καταρτήσουμε και φύλλο πορείας διότι δεν έχουμε συνολικά στατιστικά στοιχεία, αλλά ούτε και διαφοροποιημένα. Υπάρχουν κάποιε αναλύσει, αλλά μερικού χαρακτήρα, και ίσως να μην χρησιμοποιούμε και αρκετά, να μην αξιοποιούμε αρκετά το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Ίσως χρειάζεται εδώ συγκεκριμένη εντολή για διερεύνηση αυτών των θεμάτων που να απευθύνεται ακριβώς στο Ίδρυμα, στο Ινστιτούτο μας που θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να καταρτήσουμε θετικούς, ε, θετικά φύλλα πορείας. Εδώ σημείωσα με ικανοποίηση την χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για σκοπούς ε, εργασιακής ε, ένταξης των γυναικών. Βεβαίως, θα μπορούσε να είναι ένας βασικός μοχλός αυτός, ένας βασικός άξονας. Όπως είπα, ε, είναι η συμπερίληψη των νέων και των γυναικών οι δύο βασικοί άξονες που θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν εδώ. Έχετε δίκιο να τον αναφέρετε. Ε, επειδή ετοιμάζω και την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ίσως πραγματικά να μην έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτή την έκθεση στο συγκεκριμένο θέμα. Όμως ε, στην επόμενη εξέταση του θέματος πραγματικά θα κοιτάξω να επιμείνω και σε αυτό. Καλά κάνατε και μου το επισημάνατε. Θα ξαναδιαβάσω καλά το μάθημα αυτό. Επίσης σημείωσα με προσοχή την παρατήρησή σας και το πώς αναλύεται το θέμα των ε, κοινωνικών παραγόντων προστασίας. τι το χειροπιαστό έχουμε για το θέμα αυτό. Λίγα πράγματα. Όντως, σημειώνω και την ε, παρατήρηση της κυρίας Απαδοπούλου για την ε, γενιά αυτή που χάθηκε και την διαρροή ε, εγκεφάλων. Να προσέξουμε πώς θα το διατυπώσουμε, γιατί υπάρχει μια σαφής, υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός του δυναμικού ε, στις ε, διάφορες χώρες. Πρόεδρε, εντάχει αυτά ήταν όσα θεώρησα τα πλέον σημαντικά από τη συζήτηση και θα κοιτάξω τα νέα αυτά δεδομένα να τα καλύψω στην επόμενη εκδοχή της έκθεσης και να προτείνω και συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. αφήνουμε το θέμα αυτό, αφού πρώτα ανακοινώσω το χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα ψηφίσει 19 Φεβρουαρίου και θα πάει στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Έτσι μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι ο απολογισμός της ε, Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Φέμερ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας 29 με 30 Νοεμβρίου. Ε, συμμετείχα εγώ, η κυρία Άστριτ Λούλινγκ, η κυρία Μιδόρα Κρυβέτη, η Αγγέλικα Βέρτμαν και η Μαρία Κορνέλισεν. καθώς επίσης ε, μέλη της γραμματείας η Γιούτα Σούλτσε ο Ζόλταν Πέτο, καθώς ε, και τρεις ε, πολιτικοί σύμβουλοι, Φρανσίσκα Νέχερ από το ΕΛΚ, Βάλβο Λίντερ Νιόνστεν από του Σοσιαλδημοκράτες και ο Τόμ Φίλι από την ΑΛΔΕ. Ο στόχος του ταξιδιού στην Ιρλανδία ήταν να συναντηθούμε με τους Ιρλανδούς πριν την Προεδρία τους για να συζητήσουμε θέματα ισότητας μαζί τους. Πώς σκοπεύουν να προωθήσουν τα θέματα της ισότητας και στόχος ήταν και να μάθουμε πώς λειτουργούν τα ε, θέματα λιτότητας στην, ε, ισότητα συγγνώμη, στην Ιρλανδία. Ε, Καταρχήν, συναντηθήκαμε με την ε, Καθλίν Λίντς, ε, Υπουργό ε, Δικαιοσύνης, Ισότητας και Άμυνας, με την οποία θα συζητήσουμε και αύριο. Είχαμε μια μακρά συζήτηση μαζί της, τρίωρη ήταν η συνάντηση. Ε, το πρώτο μισάωρο ε, ε, το αφιερώσαμε σε θέματα άμβλωσης. Είχαμε επίσης ένα γεύμα εργασίας με μέλη του Κοινοβουλίου και το απόγευμα συναντηθήκαμε με δύο οι αρχές, να το πούμε έτσι, που ασχολούνται με θέματα ισότητας. Κατόπιν ε, συναντηθήκαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών της Ιρλανδίας, ε, το Συμβούλιο Μεταναστών της Ιρλανδίας ε, που επίσης βρίσκεται πίσω από την εκστρατεία «Σβήστε τα κόκκινα φώτα» που είναι κατά της πορνείας καθώς και το κέντρο ε, ε, ε, κρίσης για βιασμένες γυναίκες, καθώ και από την οργάνωση Ασφαλής Ιρλανδία. Η Ιρλανδία πρόσφατα άλλαξε την ομοθεσία της, ώστε... Μέχρι τις επόμενες εκλογές πρέπει να κατέχει κανείς τουλάχιστον το 30% γυναίκες και μάλιστα στις, στις επόμενες εκλογές ε, η ποσότητα των γυναικών θα πρέπει να ανέρχεται σε 40%. Τέλος, ε, συναντηθήκαμε με την κυρία Λουσίντα Κρέιτον, ε, που είναι Υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Ιλλανδίας. Συζητήσαμε μαζί της την Προεδρία. Ήταν πολύ ευχάριστο ταξίδι και νομίζω ότι όλοι το εκτιμήσαμε. Μάθαμε πάρα πολλά όλοι και νομίζω ότι είχαμε πολύ ε, ανοιχτές και γκάρδιες ε, συζητήσεις. Για παράδειγμα, συζητήσαμε το θέμα της αμβλώσης που ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητο θέμα στην Ιρλανδία. Ε, θέλησαν λοιπόν να ακούσουν τις απόψεις μας, να μας πούν τις δικές τους. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει νομίζω τουλάχιστον μεγαλύτερη κατανόηση ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Δίνω το λόγο εάν υπάρχει κάποιος που έχει να θέσει κάποια ερώτηση. Όχι. Ωραία. Κλείνουμε το θέμα αυτό και προχωράμε στο σημείο 7. που είναι αιτήσει παροχή ασύλου στην Ευρώπη συνδεόμενε με το φύλλο. Μια συγκριτική ανάλυση τη νομοθεσία των πολιτικών και των πρακτικών με γνώμονα τι γυναίκε σε εννέα κράτη-μέλη. θα γίνει η παρουσίαση από τις κυρίες ε, Λοντή Σουλάρ και Ντέμπορα Σίνγκερ που θα μας ε, μιλήσουν για τη μελέτη αυτή που έχει γίνει. Δεν ε, θέλω να μακρηγορήσω, να τους δώσω το λόγο για να μας μιλήσουν για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Παρακαλώ, καθίστε. So, please, you have the floor. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yeah, that's fine. Yeah, uh, good afternoon. Um, my... Καλό απόγευμα. Λέγομαι Ελοντή Σουλάρ. Ε, είμαι ο υπάλληλο που ασχολείται με θέματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση France d'Azil. Ε, και βρίσκεται μαζί μου εδώ η Ντέμπορα Σίνγκερ από ε, αντίστοιχη Βρετανική οργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΦΕΜ e που μας κάλεσε να παρουσιάσουμε την ε, μελέτη αυτή για αιτήσει παροχή ασύλου συνδεόμενε με το φύλλο. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω την βάση για τις ε, ευρωπαϊκές ε, συγκριτικές έρευνες που έχουν γίνει και η Τέπορα θα μας παρουσιάσει τις ε, συστάσεις μας. Καταρχήν, λοιπόν, η έκθεση αυτή ήταν μέρος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, το πρόγραμμα Jensen. Είχε διάρκεια από το 2010 μέχρι το 2012 και στόχο είχε να αυξήσει την ευαισθησία, την ε, ε, ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα θέματα ε, φύλου. Συμμετείχαν οι δύο οργανώσεις μας, αλλά επίσης και η Ισπανική, η Ιταλική και Ουγγρική μη κυβερνητική οργάνωση. Προτού να σας παρουσιάσω τα ευρήματά μας, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεθοδολογία των ερευνών. Επικεντρωθήκαμε σε εννέα χώρες ε, είχαμε ισορροπία ανάμεσα στις βόρειες, νότιες, ανατολικές και δυτικές χώρες, ε, καθώς και ανάμεσα σε χώρες που ε, δέχονται μεγάλο ή μικρό αριθμό ετούντων ασύλου. Άσυλο. ήταν ποιοτική και ποσοτική έρευνα. συλλέξαμε 132 ερωτηματολόγια από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων ασχοληθήκαμε με πολιτικές, νομοθεσία, πρακτικές ε, όσον αφορά το καθορισμό του καθεστώτος, ε, τις ε, διαδικασίες και την κράτηση των γυναικών ετούν τον άσυλο. Επίσης είχαμε 60 συνεντεύξεις με γυναίκες που ζητούν άσυλο ή που είναι πρόσφυγες στις χώρες αυτές τα βασικά μας ευρήματα. Αν κοιτάξουμε τις στατιστικές, ε, βλέπουμε ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο των ετούντων άσυλο στην Ευρώπη κατά μέσο όρο. Ωστόσο, Υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ ανάμεσα στι διάφορε χώρε. Για παράδειγμα, η Σουηδία και η Γαλλία δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών ετούν τον άσυλο, ενώ η Ουγγαρία και η Ιταλία δέχονται τον ε, μικρότερο αριθμό αιτήσεων. Επίσης, ε, το ποσοστό ε, αναγνώρισης ε, όταν αναλυθεί ανάλογα με το φύλλο, βλέπουμε ότι αποκαλύπτει διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και μιλάμε για καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς προστασίας. Ε, όσον αφορά τις στατιστικές, θα θέλαμε να τονίσουμε μια καλή πρακτική που ε, παρατηρήσαμε στο Βέλγιο. Ε, είναι η μόνη χώρα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένε στατιστικέ όσον αφορά ε, τι αιτήσει ασύλου αναλυμένε ε, αναφύλω. Ε, εφτά είδη ε, αιτήσεων ε, για άσυλο που συνδέονται με το φύλλο έχουν εντοπιστεί. Δεν είναι εξαιρετικός ο κατάλογος, αλλά δίνει μια ιδέα σχετικά με τις αιτίες για, την, για τις αιτήσει ασύλου. Βλέπουμε ότι διάφορες χώρες έχουν αναπτύξει κατευθυντήρες γραμμές ε, για, τους, ε, για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και που γενικά ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήρες γραμμές ε, για το φύλλο του, της υψηλής αρμοστίας προσφύγων του ΟΗΕ. Στόχο έχουν εναρμόνιση των αιτήσεων ασύλου σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ χρήσιμες οι κατευθυντήρες γραμμές αυτές για το προσωπικό, αλλά ο αντίκτυπός τους είναι κάπως περιορισμένος στην πράξη, διότι είναι ένα μη δεσμευτικό έγγραφο. Οι έρευνες ε, επικεντρώθηκαν ε, στον καθορισμό του καθεστώτος. Ε, εξετάσαμε δηλαδή πώς τα θέματα φύλου ερμηνεύονται στο νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Γενέβης ε, καθώς ε, και την σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενέβης, μπορεί να δοθεί καθεστώς πρόσφυγα σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει βάσιμους λόγους να φοβάται δίωξη για λόγους θρησκευτικούς, εθνοτικούς κτλ. και που βρίσκεται εκτός της χώρας προέλευσής τους και λόγω του φόβου του δεν ε, θέλει να προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό αυτών, Μελετήσαμε σε τι βαθμό η βία λόγω φύλου ε, θεωρήθηκε δίωξη, σε τι βαθμό τα, οι όροι αυτοί του ορισμού ε, ερμηνεύονται ε, ανάλογα με το φύλλο και ε, κατά πόσο οι διαδικασίες ε, θεωρούνται αξιόπιστες. Ε, διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες κακές πρακτικές όσον αφορά την ερμηνεία της βίας λόγω Για παράδειγμα στη Γαλλία δεν θεώρησαν την οικιακή βία ή τον βιασμό και την σεξουαλική βία ως δίωξη και επίσης στην Ισπανία ε, δεν θεωρούν ότι ε, η εμπορία ανθρώπων θεωρείται δίωξη και γι' αυτό οι γυναίκες που ζητούσαν άσυλο για τους λόγους αυτούς δεν μπόρεσαν να λάβουν ε, καθεστώς πρόσφυγα. Όσον αφορά τους λόγους για την παροχή ασύλου, οι έρευνες δείχνουν ότι η Ρουμανία είναι η μόνη χώρα που έχει προσθέσει το φύλλο ως ε, επιπλέον ε, λόγο για την παροχή ασύλου. Αυτή είναι καλή ε, πρακτική, διότι ούτε η Σύμβαση της Γενέβης, ούτε η σχετική οδηγία θεωρεί ότι αυτός είναι ξεχωριστό λόγος για την παροχή ασύλου. Επίσης, όσον αφορά την ερμηνεία των όρων, των προϋποθέσεων που αναφέρονται στον ορισμό, δείχνει ότι γίνεται δυσανάλογη ερμηνεία και μάλιστα άσχετα από τις συστάσεις της ΥΠΑ ε, της Αρμοστίας να ερμηνεύονται και οι πέντε προϋποθέσεις ε, με λόγο που να αντικατοπτρίζουν και το φύλλο. Ιδιαίτερα ε, όταν μιλάμε για θρησκευτικούς λόγους. Ε, Επίση ε, προβληματικό είναι ότι οι αιτήσει παροχή ασύλου που συνδέονται με το φύλλο ε, εξετάζονται με βάση την κοινωνική ομάδα. Υπάρχει πολύ διαφορετική ερμηνεία ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη πάνω στο θέμα αυτό. Κάποια κράτη-μέλη επικαλούνται τον ορισμό αυτό, ότι το φύλλο μπορεί να είναι λόγος για την συμμετοχή σε κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ενώ η Γαλλία ερμηνεύει πιο ε, περιοριστικά τον όρο αυτόν. Υπάρχει Λοιπόν, αρκετή μεγάλη διαφορά στην προστασία που δίνεται στις γυναίκες ανάλογα με τη χώρα στην οποία κάνουν την αίτηση ασύλου. Πολύ σημαντικό θέμα στον ορισμό του πρόσφυγα είναι το θέμα των βάσιμων φόβων δίωξης. Πρέπει δηλαδή να θεωρηθεί αξιόπιστη, ε, αξιόπιστος ο φόβος και όσον αφορά τις ε, αιτήσει ασύλου που συνδέονται με το φύλλο, το θέμα αυτό είναι πολύ προβληματικό διότι πολύ συχνά οι γυναίκες δυσκολεύονται να μιλήσουν για τους φόβους τους. Ε, επειδή ενδεχομένω εμπλέκονται μέλη ε, οικογενειακά, φοβούνται Μπορεί να φοβούνται, μπορεί να ντρέπονται, μπορεί να ε, ε, ε, νιώθουν τραυματισμένες και γι' αυτό διστάζουν να αποκαλύψουν τις σχετικές πληροφορίες. Η αξιοπιστία λοιπόν είναι σημαντικός λόγος απόρριψης των αιτήσεων. Οι γυναίκες θεωρούν ότι η βία που οφείλεται στο φύλλο δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, διότι τι τεκμηρίωση μπορεί να υπάρξει ε, σε περίπτωση βιασμού ή οικιακής βίας. Πόσο μάλλον σε περιπτώσει όπου δεν είναι δυνατόν να προσφύγει κανεί στην αστυνομία στη χώρα προέλευση. Έτσι λοιπόν οι γυναίκε ε, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Οι έρευνε δείχνουν ότι γενικά οι χώρε ε, δυσκολεύονται να λάβουν υπόψη του τι δυσκολίε αυτέ κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλου. Και πολύ συχνά δεν, δεν πιστεύουν οι αρχέ τι γυναίκε. Ε, θα περάσω κάπως γρήγορα κάποιες διαφάνειες. Όπως ε, μόλις είπα λοιπόν, οι γυναίκες ε, που φοβούνται την δίωξη που οφείλεται στο φύλλο, φοβούνται να μιλήσουν για τις φοβίες τους, για τους φόβους τους και κάποιες γυναίκες μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι μπορούν να ζητήσουν άσυλο για λόγους που έχουν να κάνουν με το φύλλο. Ε, θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν κάποια διαδικαστικά έργα ε, στα διάφορα κράτη-μέλη, όπως είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες, ε, τα χρονοδιαγράμματα, η διαπίστωση συγκεκριμένων αναγκών και να γίνονται και συνεντεύξει. Επίσης, να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα καλής πρακτικής ε, στο Βέλγιο. Έχει εκδώσει ένα φυλάδιο που λέγεται «Γυναίκες και ε, κορίτσια που ζητούν ε, άσυλο στο Βέλγιο». Έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και παρέχει πληροφορίες για κάποια θέματα όπως είναι η εγκυμοσύνη, η αντισύλληψη, η υγεία, ε, η οικιακή βία και η εμπορία γυναικών. Είναι η μόνη χώρα όπου η αρμόδια αρχή ε, παρέχει τις πληροφορίες σε γυναίκες που ζητούν άσυλο. Έχουμε εντοπίσει όμως και κάποιες κακές πρακτικές, όπως για παράδειγμα ενώ η επιταχυμένη διαδικασία ασύλου μπορεί να εμποδίσει τις γυναίκες να αποκαλύψουν ε, πληροφορίες, είδαμε ότι ε, καμία χώρα δεν ε, απέκλειε τις αιτήσει ασύλου λόγω φύλου από τις κανονικές διαδικασίες ρουτίνας. Επίσης, ε, σημαντικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση της αίτηση ε, είναι ότι ε, ο ετών θα πρέπει να μπορεί προφορικά να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την συνέντευξή του. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την δυνατότητα μιας γυναίκας να αποκαλύψει πληροφορίες, για παράδειγμα, το φύλλο του συνομιλητή ή του διερμηνέα κατά τη συνέντευξη, καθώς και η παρουσία των παιδιών τους στο δωμάτιο. Δεν θα μπω σε αναλυτικέ λεπτομέρειε, αλλά οι έρευνε δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιε καλέ πρακτικέ, ιδιαίτερα σε βόρειε χώρε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και το Βέλγιο. όσον αφορά την εκπαίδευση. Παρά ε, τα παραδείγματα καλών πρακτικών σε κάποιες ε, χώρες υπάρχει έλλειψη κατάρτισης ε, το, αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις. Γενικά είδαμε ότι οι αρχές ασύλου δεν καταλαβαίνουν και δεν αντιμετωπίζουν θέματα που έχουν να κάνουν με το φύλλο κατά τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος. Μετά λοιπόν από τα διαδικαστικά θέματα, οι έρευνες μας ε, επικεντρώθηκαν και σε, ε, στις συνθήκες υποδοχής των γυναικών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε και πάλι, αλλά τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά. Ε, βρήκαμε διάφορες αναφορές περιστατικών βίασης βάρος γυναικών ε, που ζητούν άσυλο, ε, ιδιαίτερα ε, σεξουαλικές επιθέσεις σε μη συνοδευόμενες γυναίκες ή οικιακή βία σε περιπτώσεις γυναικών που συνοδεύονται από τον σύντροφό τους όταν αντιμετωπίζουν βία που οφείλεται στο φύλλο είναι τελείως αβοήθητες στη χώρα ασύλου. Θα ήθελα να τονίσω Ένα θέμα που έχει να κάνει με τις ε, άσυλο που ε, με τους ετούντες άσυλο που τραπετεύουν ε, από τα δίκτυα εμπορίας. Χρειάζονται ασφαλή μέρη παραμονής και μόνο στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε ότι υπάρχουν ειδικά κέντρα υποδοχής για ετούντες άσυλο θύματα εμπορίας. Σε κάποιες άλλες χώρες ε, μπορεί να υπήρχαν ε, ε, μέρη στέγασης των θυμάτων εμπορίας, δεν ήταν προσαρμοσμένα όμως και για το άσυλο. Τέλος, όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, ε, είναι πολύ κακές ε, για όλους τους ετούντες άσυλο στην Ευρώπη, αλλά οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Για παράδειγμα, οι ασυνόδευτες γυναίκες ε, όταν περιστοιχίζονται από, από άγαμους άντρες ή γυναίκες με παιδιά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Και πάλι υπάρχει πρόβλημα έλλειψης κατάρτισης του προσωπικού στα κέντρα κράτησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνε δείχνουν λοιπόν ότι παρότι έχουν εντοπιστεί κάποιε καλέ πρακτικέ σε κάποιε χώρε, ε, η μεταχείριση των γυναικών που ζητούν άσυλο δεν ε, έχει προσαρμοστεί στην. Ε, δεν έχει υποστεί προσαρμογές στην πράξη. So, what are the implications of these? Ποιε είναι οι επιπτώσει από τα ευρήματα αυτά για τις γυναίκες που δούνται άσυλο και ποιε είναι οι δικέ μας τι στάσει. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των χωρών όπου έγινε η έρευνα και ασυνέπειες, χαμηλά πρότυπα και πολύ κακή υλοποίηση των πολιτικών όπου υπάρχουν. Για να σας δώσω κάποια παραδείγματα αυτών των καλών και κακών πρακτικών, τι θα γίνει στο Βέλγιο αν μια γυναίκα έτυχε άσυλο μπορεί να τη δοθεί ένα φυλάδιο που διατίθεται σε 7 διαφορετικέ γλώσσε για την ισότητα των φύλων, αλλά στη Μάλτα θα πρέπει να, ε, να αποφασίσει αρμόδια υπηρεσία για την ε, πρώτη εκδίκαση για την ε, αποδοχή μάλλον της αίτησης ή ένα δικαστήριο με έφεση. Στη Γαλλία μπορεί κανείς να στεγαστεί σε ένα κέντρο για αστέγους. Αλλά αυτό που λένε οι γυναίκε είναι ότι δέχονται πιέσει για να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με άντρε χωρί να μπορούν να καλέσουν την αστυνομία. Υπάρχει η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα στις Ισπανικές, στην Ισπανία όμω, οι αρχέ δεν θεωρούν ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί αδίκημα. Δεν το αναγνωρίζουν. Έτσι λοιπόν, πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαζόταν πολιτική για την αποδοχή επίσης ασύλου, όμως περισσότερες ε, χώρες δεν διαθέτουν κάτι τέτοιο. Η Σουηδία βλέπουμε ότι ακολουθεί διαφορετική πρακτική από ό,τι άλλες χώρες και πολλές φορές είναι οι πολιτικοί που ερμηνεύουν την ε, δημόσια γνώμη. Όπως ε, το τι γίνεται στην Βρετανία με διάφορες περιφέρειες που προσφέρουν και περίθαλψη για τα παιδιά κατά την συνέντευξη για την ε, αίτηση ασύλου. Όμω, όταν κανείς λάβει την επίσημη αίτηση, βλέπει ότι λέει μη φέρτε τα παιδιά σας γιατί δεν παρέχετε πρόνοια για τα παιδιά. Στην Ουγγαρία τώρα, οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες και μπορεί να βρεθούν σε κράτηση ή, στην Ιταλία όπου υπάρχει κράτηση αλλά χωρίς την παρακολούθηση μάλλον στην ε, Ιταλία υπάρχει παρακολούθηση από γιατρό και αρμόδιες υπηρεσίες Βλέπουμε η νομοθεσία για την αποδοχή αιτήσεων ασύλου από γυναίκε που είναι και θύματα ενδοοικογενειακή βία δεν έχει προσαρμοστεί. Δεν χρειάζεται να ε, είναι μεγάλη προσπάθεια των κρατών που διαθέτουν τέτοια πολιτική αρκεί να δουν τα κοινωνικά κράτη και τις καλές τους πρακτικές. Η Ελλοντία από τη γαλλική Τέντα δείχνει ποια είναι τα κενά ε, της γαλλικής νομοθεσίας. Γι' αυτό και διοργάνωσε μια επίσκεψη μελέτης από την Βρετανία ε, προς, το, προς τη γαλλική υπηρεσία. Υπήρξε ανταλλαγή λοιπόν ε, στοιχείων και από τις δύο πλευρές ώστε να γίνει καλή ανταλλαγή, ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αυτό θα μπορούσε να γενικευθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να είμαστε όμω ανεκτικοί με τι χώρε που διαθέτουν καμία πολιτική. Θα πρέπει τα συστήματα αποδοχή αιτήσεων ασύλου να λαμβάνουν υπόψη και το φύλλο, όμω ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε για το σκοπό αυτό. Μετά από μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο Παρίσι το Σεπτέμβριο του 2011, όπου συμμετείχε η κυρία Λάμπερτ, και άλλοι νομικοί, ειδικοί, μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ε, εκπρόσωποι της ε, είπα της Δικαιώματα του ΙΕ ε, συζητήθηκαν εκεί τα ερευνητικά πορίσματα ώστε να καταρτήσουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να λάβουμε. Η Τζιν Λάμπερτ οργάνωσε συνάντηση για να ξεκινήσει η έκθεση η εξέταση της έκθεσης αυτής στο Κοινοβούλιο το Μάιο του 2012. Σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα που επανεκδώσατε την έκθεση αυτή τώρα από την Επιτροπή των Γυναικών και να σα απευθύνουμε τι βασικέ μα συστάσει. Αυτέ είναι οι προτεραιότητέ μα. Πρώτα απ' όλα, τα επιμέρου κράτη-μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν κατευθυντήριε γραμμέ για τα φύλλα, ώστε να ε, γνωστοποιηθούν αυτέ και στου δικαστέ και να βασιστούν στι κατευθυντήριε γραμμέ τη υπό τη Αρμοστία του ΙΕ. Εφόσον εγκριθούν οι γραμμέ αυτέ, θα πρέπει επιπλέον να ε, υλοποιούνται κιόλα. Επίση, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όπω τα ξέρετε, η Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για τη Βία κατά των Γυναικών, κατά πολέμηση τη βία κατά των γυναικών, έχει ένα πολύ έντονο άρθρο για τα θέματα ασύλου. Θα πρέπει, όπω και το Ευρωκοινοβούλιο, όπω και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνουν την ισότητα το φύλλο μάλλον στην κατάρτιση και το σχεδιασμό πολιτικών και οι πολιτικές αυτές όντως να υλοποιούνται. Διότι αν οι ανάγκες και τα δικαιώματα των γυναικών που δούνται άσυλο αγνοούνται συστηματικά, αυτό αποτελεί ένα πραγματικό κενό. Το 2010 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε έκθεση για τις ε, προσφυγές ε, που σχετίζονται με θέματα ασύλου από γυναίκες. Εδώ χρειάζεται να δημιουργηθούν συστήματα ασύλου ευαίσθητα ω προ τη διάσταση του φύλου σε όλα τα κάτι μέλη. Αυτό κατέδειξε η σχετική μελέτη. Οι συστάσει για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίω για την ΓΙΑΖΟ, που είναι η υπηρεσία στήριξης των συστημάτων ασύλου, είναι σημαντικό να αναλάβουν εδώ ρόλο. Πρέπει να ισχύει αυτό ακόμη και για τους ε, πολίτες τρίτων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε σε αυτό το δίκτυο το συμβουλευτικό συστάσεις ώστε να λάβει υπόψη την ισότητα των φίλων σε όλες τις διαστάσεις των εργασιών του και στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Την συλλογή επίσης πρωτότυπων και ε, επί της πράξης ε, πληροφοριών και ιδίως από τα συστήματα εξέτασης αιτήσεων ασύλου των κρατών μελών. Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε ότι το πρόγραμμα εργασιών του 2013 της ΙΑΖΟ αναφέρεται στα θέματα ε, του φύλου και στην εκπαίδευση και στην περίπτωση του ελέγχου της ποιότητας. Και στην ΙΑΖΟ και στο Ευρωκοινοβούλιο ελπίζουμε ότι θα παρακολουθείτε την πρόοδο στα θέματα ισότητας των φύλων οι συστάσει μα όμω δεν απευθύνονται μόνο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Πιστεύουμε ότι είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ ε, θα πρέπει να περιλάβει ένα σύνολο προτεραιοτήτων που να σχετίζονται με την ισότητα των φύλων για όλου του ευθύνοντε και λαμβάνοντε αποφάσει σε υψηλά κλιμάκια. Και αυτά να είναι εύκολα προσβάσιμα και στι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Το ίδιο και για όσου ξεκινούν εκπαίδευση και καταρτίζουν σχετικά προγράμματα. Αυτό φάνηκε ότι καλό είναι να προωθηθεί ω ιδέα γιατί υπάρχουν και δυνατότητε άσκησης πίεσης. Πολλές φορές οι γυναίκες που τον άσυλο είναι θύματα εμπόρων, διακινητών και είναι απελπισμένες ε, υπολογίζουν στην τύχη τους, ε, την καλή του τύχη, αλλά πολλέ φορές πέφτουν θύματα κακής μεταχείρισης. Για σκοπούς λοιπόν ε, συνοχής θα πρέπει να αυξήσουμε τα σχετικά πρότυπα. Θα πρέπει κάθε γυναίκα να μπορεί να προστατεύεται από κάθε είδου δίωξη σε οποιοδήποτε κράτο μέλο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σουηδικά θα μιλήσω, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποια σύντομη ερώτηση. Όχι. Θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη σας. Και υπάρχουν πολλά θέματα από αυτά που αναφέρατε με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί κανείς. Είναι απίστευτες οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν άμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. υπάρχουν καλές πρακτικές. Και υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουμε τις βέλτιστες αυτές τις πρακτικές, να πούμε ότι υπάρχει εδώ ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, οι συστάσεις που μας κάνατε, που είναι εύκολο να τις υιοθετήσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχει βέβαια αποφασίσει ακόμα η ε, Επιτροπή μας, αλλά θα, μπορούσαμε, θα μπορούσαν τα θέματα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ε, έκθεσης πρωτοβουλίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να εκμεταλλευτούμε το υλικό που υπάρχει στην έκθεσή σας, ε, διότι υπάρχουν πολλά χρήσιμα πράγματα σε αυτήν. Η κυρία Κώστα ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ, ε, αλλά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να εκφράσω την εκτίμησή μου για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ξέρω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Όμως συμφωνώ απολύτως με σας, Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα ζήτημα όπου καλό θα ήταν να αναλάβει μια έκθεση πρωτοβουλίας ε, η Επιτροπή Γυναικών. Αφορά τη δέσμη μέτρων για το άσυλο γενικότερα. Το να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στη διάσταση των φύλων, στο πλαίσιο των πρακτικών και εθνικών νομοθεσιών, είναι νομίζω κέρια σημασίας. Τη μελέτη βέβαια αυτή πρέπει να τη διαβάσει κανείς και να τη μελετήσει με προσοχή. Διότι υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Όταν μιλάτε για τόσο διαφορετικές περιπτώσεις και μιλάτε για καλές πρακτικές που ισχύουν σε διαφορετικές μεταξύ τους χώρες, ε, είδαμε τι γίνεται σε χώρες του Βορρά, αλλά και στην Ιταλία, τη δική μου χώρα, πολλές φορές έχουμε παραδείγματα, εγώ τη γνωρίζω εκ του σύναγκη στην ε, κατάσταση αυτή, αλλά ξέρω τι γίνεται με τις γυναίκες που είναι πρόσφυγες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, συγκεκριμένες καλές πρακτικές υποδοχής και θα μπορούσε να οργανωθεί ένα σεμινάριο για να αφηγηθούμε και με λεπτομέρειες τις καλές αυτές πρακτικές. Θα σταματήσω εδώ, υπόσχομαι να μελετήσω, να διαβάσω με προσοχή την έκθεση αυτή αλλά η γνώση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των φορέων τοπικής αυτοδίκησης, καθώς και τα δικά σας ε, στοιχεία και παρατηρήσεις, νομίζω ότι μπορούν να, δώσουν, να ρίξουν φως μια διάσταση του θέματος που πολύ συχνά δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη. Ωραία, θέλετε να κάνετε κάποια τελευταία παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ακούω την ίδια μου τη φωνή. Ε, ευχαριστώ για αυτή την τόσο θετική αντίδραση. Η έκθεση βρίσκεται εδώ. Είναι πια δική σας έκθεση και στα αγγλικά ε, και στα γαλλικά, χάρη στην Ελλοντή. Δυστυχώς όχι στα ταλικά, λυπάμαι γι' αυτό αλλά πραγματικά μας απασχόλησε να μην πούμε ότι σε μια χώρα κάνουν μόνο στραβά ή σωστά. Όλες οι χώρες μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους ε, θετικά στοιχεία και εμπειρίες. Υπάρχουν παραδείγματα καλών πρακτικών παντού. Είναι λοιπόν εύκολο να γίνει ανταλλαγή. Εάν ήταν όλα μαύρα, δεν θα ξέρουμε πού να αρχίσουμε. Αλλά το να πούμε αυτό το καλό γίνεται στην Ιταλία, στη Μάλτα ή στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πιο απλό εύκολα μπορεί να επιταχυνθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που ήρθατε εδώ σήμερα. Eh, Ωραία. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Και προχωράμε στο τελευταίο σημερινό θέμα, το υπαριθμόν 8. Επίσκεψη μελέτης για γυναίκες βουλευτές της Νοτίου Συνισταμένης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι στο κανάλι 21 υπάρχει διερμηνία στα αραβικά. Ελπίζω να βρήκατε το σωστό κανάλι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τις γυναίκες βουλευτές από την Τινησία, τη Λιβύη και το Μαρόκο. Σας καλωσορίζω θερμά. Χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε εδώ. Ήρθατε για να δείτε πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο μας. Και μάλιστα είναι πολύ επίκαιρη η επισκέψη σας για τις δικές μας εργασίες. Ε, διότι έχουμε και εμείς τη δική μας επίσκεψη στην Τινησία. Βέβαια, ε, δεν ε, έχουμε χρόνο για περισσότερες χώρες, αλλά ε, θα εκπονήσουμε έκθεση πρωτοβουλίας ε, που θα ψηφιστεί την επόμενη, ε, τον επόμενο μήνα. Ε, χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία να μας μιλήσετε για τη δουλειά σας. Αλλά πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κώστα, που είναι η συγγήτρια για την έκθεση «Γυναίκες στη Βόρεια Αφρική». θα αναφερθεί στα θέματα που εξετάζει η έκθεσή της και κατόπιν θα έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε γιατί βρίσκεστε εδώ και να μας μιλήσετε για τη δικιά σας δουλειά. Η κυρία Κώστα πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπάμαι που έχω γυρισμένη την πλάτη στις προσκεκλημένες μας που βρίσκονται στο βάθος της αίθουσας αλλά δυστυχώς έτσι είναι η χωροταξία της αίθουσας. Νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία και για μας είναι συγκινητικό επίσης και πολύ ευχάριστο όχι μόνο για μένα, για όλες τις συναδέλφους, να μπορούμε να φιλοξενήσουμε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση. Όπως έλεγε προηγουμένως ο πρόεδρος Γκούσταυσον, ως Επιτροπή Γυναικών θελήσαμε να συντάξουμε έκθεση πρωτοβουλίας από πλευράς της Επιτροπής μας για την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική, συγκεκριμένα σε τέσσερις χώρες που λάβαμε υπόψη στην εκθέση αυτή, τη Λιβύη, την, την Ισία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο. Σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε εδώ βουλευτές από τη Λιβύη, την Τινησία, το Μαρόκο και ίσως να μην ήρθαν γυναίκες από την Αλγερία. Δεν ξέρω αν κατάφεραν να φτάσουν. Γνωρίζετε. Μάλιστα, όντω δεν κατάφεραν να φτάσουν. Και νομίζω δεν υπάρχουν βουλευτές από την Αίγυπτο. Αυτό που θέλαμε κυρίως να εξετάσουμε είναι η κατάσταση των γυναικών που συμμετείχαν οι ίδιες αυτοπροσώπως ε, στην διαδικασία που ονομάζεται και Αραβική Άνοιξη στις χώρες αυτές. Σήμερα γνωρίζουμε ότι παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες, πολλές δυνατότητες χάρη σε αυτό το φαινόμενο, πολιτικές διαδικασίες που βρίσκονται ακόμα να εξελίξει, αλλά και κάποιες καταστάσεις ε, σύγκρουσης που ανησυχούν. Πράγματι, η κατάσταση των γυναικών, καθώς και το κατά πόσον ανέλαβαν οι γυναίκες πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι σημαντικό. Όπω επίση και το πώ αποτιμάται όλη αυτή η κατάσταση στην Τινησία, με την επίσκεψή μα, ε, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε από τα δικά σα τα λόγια, τι δικέ σα τι διηγήσει, την διαδικασία, την δημοκρατική ε, εξέλιξη στι χώρε αυτέ και το κατά πόσον προωθούνται τα δικαιώματα και οι ανάγκες των γυναικών, κατά πόσον δόθηκε δηλαδή και μια εξουσία, ένα κύρος στις γυναίκες και τη θέση τους. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί της έκθεσής μου. Ε, ιδιαιτέρως ε, προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε σε τέσσερις πτυχές της ε, σημερινής κατάστασης. Πρώτον, να θυμίσουμε και να αναγνωρίσουμε, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε των τεσσάρων χωρών που εξετάστηκαν, πώ συμμετείχαν οι γυναίκε στι επαναστατικέ διαδικασίε τη βαθιά αυτή μεταβολή και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, των εκλογών μάλλον που διοργανώθηκαν ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκαν ελεύθερε εκλογέ λόγω χάρη στη Λιβύη. Ένα πρωτοφανέ πολιτικό φαινόμενο με ανάλογο αντίκτυπο. Και στην Τινησία νομίζω 27% των εκλεγμένων ήταν γυναίκε. Και ε, συμμετέχουν στις επιτροπέ που εξετάζουν την συνταγματική μεταρρύθμιση της Τινησία. Και στη Λιβύη όμως βλέπουμε μια πραγματική καινοτομία. 17% γυναικών στο κογκρέσο της χώρας ή στην ε, Αίγυπτο όπου υπήρξε μείωση της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογές διότι δεν υπήρξε εκλογικός νόμος που να τις ευνοεί, να τις καλύπτει με κάποιες ποσοστώσεις. Παρόλο λοιπόν που είναι εύρωστη, ευρωστότατη η κοινωνία των πολιτών ε, και τα κοινωνικά δίκτυα στην Αίγυπτο, στο Μαρόκο η μεταρρύθμιση είχε ήδη ξεκινήσει και νομίζω οι γυναίκες συμμετείχαν ήδη ενεργά στις περισσότερου φορείς. Το πρώτο λοιπόν σημείο ήταν να φανεί ε, με γλαφυρότητα το στοιχείο της συμμετοχής των γυναικών, ακούγοντας και τις δικές σας εμπειρίες, τις δικές σας μαρτυρίες, καθώς είστε βουλευτές και θέλαμε να γνωρίζουμε πώς εξελίχθησαν τα γεγονότα στις χώρες σας. Ιδίω ό,τι αφορά την συμμετοχή σε κοινοβουλευτικά σώματα, αλλά και κάτι στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση. Πώς δημιουργούνται ε, δυνατότητες στήριξης για την κοινωνία των πολιτών, τις ενώσεις γυναικών, τις οργανώσεις γυναικών, ώστε να στηριχθεί το δικό σας το έργο. Και με την δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων και με τις νέες νομοθεσίες για τα δικαιώματα των γυναικών. Ακούσαμε ότι ένα από τα σοβαρότατα αιτήματα ε, και στην Τινησία και στην Αίγυπτο είχαμε πολλές τέτοιες συναντήσεις, ακροάσεις. Ήταν να προβλεφθεί στο Σύνταγμα η ισότητα των γυναικών και της προστασίας των δικαιώματων των γυναικών, να ε, υλοποιηθούν οι διεθνείς συμβάσεις, ιδίως για το άσυλο αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τις γυναίκες, ώστε να κατοχυρώνονται και τα δικαιώματά τους μεταξύ των οικουμενικών θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εδώ ήθελα να ακούσω και τι δικέ σα απόψει, αλλά και για την δυνατότητα ε, ανάθεση εξουσία στι γυναίκε. Ε, Ποιε είναι οι αδυναμίε, ποια τα δυνατά σημεία τη θέση των γυναικών. Ε, σε πολλέ περιπτώσει ακούμε ότι στι χώρε αυτέ είναι λόγω χάρη ιδιαίτερα συχνή παρουσία γυναικών στου ακαδημαϊκούς κύκλους, αλλά όχι στι περιπτώσει τη οικονομική ανάπτυξη. Στην Τινησία όμως ε, οι γυναίκες ε, είχαν ενεργότερο ρόλο από ό,τι σήμερα που έχουν ξεκινήσει και διαφωνίες με κάποιες ε, περιπτώσεις παλινδρόμησης. Έτσι λοιπόν και σε σχέση με τις οικονομικές δυσχερίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές θα θέλαμε να καταλάβουμε αν οι γυναίκες υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν σε θέση περιθωριακή, περιθωριοποίησης να ακούσουμε πάλι και για αυτό το θέμα τις δικές σας απόψεις. Και τρίτο σημείο, εξαιρετικά σημαντικό, η δική μας ευθύνη, και ολοκληρώνω εδώ, η δική μας ευθύνη ως Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι γνωρίζετε ότι διαθέτουμε διαφορετικά μέσα, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί, χάρη στη νέα πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, την, με τις χώρες της Μεσογείου, και αυτό επιτρέπει πρωτοβουλίες και διμερείς και περιφερειακές και πολυμερείς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μάλλον περισσότερα και εδώ θέλω περισσότερες ιδέες, προτάσεις από εσά, ώστε οι γυναίκες να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με αυτά τα προγράμματα συνεργασίας. Διότι υπάρχει και η ε, προοπτική του More for More και ε, θέλουμε βέβαια να προχωρήσει η διαδικασία δημοκρατισμού στις χώρες αυτές, αλλά ε, να κατοχυρωθεί και η θέση των γυναικών σε όλη αυτή τη διαδικασία και η προστασία των δικαιωμάτων τους. Ε, ελπίζω να καταλαβαίνουν οι βουλευτές που είναι σήμερα μαζί μας ότι μπορούν να μας θεωρούν συμμάχους. Εγώ στηρίζω τις δικές τους ε, προσπάθειες, τους δικούς τους αγώνες και από αυτή την προοπτική ήθελα να καταλάβω και ποιες είναι οι δικές τους οι προτεραιότητες. Στον κατάλογο των προτεραιοτήτων που θεωρούν ότι θα μπορούσε να ενισχύσει η Ευρώπη τις δικές τους τις επιδιώξεις, ε, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα στοιχεία και να δούμε ποια είναι τα κομβικά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Εδώ θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει διάλογος πολυκομματικός των γυναικών που βρισκόμαστε εδώ, ώστε να προωθήσουμε κοινού στόχου. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. Νομίζω ότι έχετε θέσει πολύ καλά ερωτήματα, στα οποία θα ήθελα και εγώ να ακούσω απαντήσεις. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά μήπως είναι δυνατόν ε, τουλάχιστον μία από κάθε χώρα να πει λίγα λόγια. Πέντε λεπτά τη διάθεσή σας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Αποφασίστε εσείς ποια θα ξεκινήσει. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ε, καλώς ορίσατε θερμά. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Εγώ είμαι μέλος ε, της Βουλής της Τινησίας και θα ήθελα να μιλήσω στα αραβικά γιατί είδα ότι εδώ υπάρχει πολυγλωσία και γι' αυτό θα μου άρεσε να ακουστεί και η αραβική γλώσσα. Η κατάσταση στην Τινησία, όπως είπε και η κυρία Κώστα είναι μεταβατική. Η κυρία Κώστα το εξήγησε πάρα πολύ καλά αυτό. Κάθε μεταβατικό στάδιο, όπως γνωρίζετε, ε, χαρακτηρίζεται και από ανησυχίες και από διαφόρων ειδών ε, καταχρήσεις και από ε, παρεκκλήσεις και εκτροχιασμούς, θα έλεγα. Όλα αυτά εξηγούν το τι συμβαίνει μέσα στην Εθνική Συντακτική Συνέλευση. Βρισκόμαστε στη διαδικασία κατάρτισης του Συντάγματος σήμερα. Δεν έχουμε άλλη ανελακτική ε, λύση από την εθνική ομοψυχία, την εθνική ε, συνένεση. Πρέπει να συνενέσουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Σημειώσατε την καθυστέρηση ως προς την διοθέτηση ε, του κώδικα για το καθεστώς του προσώπου. Εμείς όμως ε, ε, θα επιμείνουμε για να μην τροποποιηθεί ο κώδικας αυτός προς τα κάτω και να μην αλλάξει το καθεστώς των ατόμων. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες όλων. Είναι ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο συγκριτικά με το Σύνταγμα του 59. Είναι και βελτίωση αυτή, σημείο στο οποίο έχουμε βελτίωση. Με το νέο κείμενο την Προεδρία μπορεί να αναλάβει και γυναίκα. Στο προηγούμενο Σύνταγμα αυτό δεν είχε αναφερθεί ρητός. Αναφέρατε επίσης ότι έχουμε νομοθετικές επιτροπές, συντακτικές επιτροπές. Πράγματι, υπάρχουν αυτές στην Εθνική Συντακτική μας Συνέλευση και παρίστανται γυναίκες στις επιτροπές αυτές. Η γυναίκα στην Τινησία λοιπόν σήμερα, έτσι όπως τη γνωρίζουμε από την εποχή των απικιών, είναι παρούσα. Η γυναίκα είναι πάντοτε παρούσα, ήταν πάντοτε παρούσα. Ε, πάρα πολλές γυναίκες ε, πηγαίνουν στο σχολείο, νεαρά κορίτσια. Το ποσοστό ε, σχολικής εκπαίδευσης των κοριτσιών στη Ισία είναι πιο υψηλό συγκριτικά με το ποσοστό των αντίστοιχων αγοριών. Αυτό συνέβαινε πάντοτε από την εποχή των απικιών μέχρι και σήμερα. Και αυτό οφείλεται πέραν της πολιτικής ε, και στην οτροπία της κοινωνίας μας. Δεν μπορεί κανείς να καταγγέλει την αραβική κοινωνία για καθυστερήσεις στον τομέα αυτό, διότι η αραβική κοινωνία μέχρι τώρα διαβιούσε υπό το καθεστώς μονοκομματισμού και δικτατορίας. Σε μια λοιπόν ε, τέτοια ε, κοινωνία η γυναίκα αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με αυτές που αντιμετωπίζουν και οι γυναίκες στη Δύση. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνδέσουμε την κατάσταση των γυναικών στη χώρα αυτή με την εμφάνιση ε, του νέου ε, Ισλαμικού κόμματος, για παράδειγμα, σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Βλέπετε ότι εγώ είμαι σύγχρονη γυναίκα, είμαι δραστήρια, ενεργή. Εξελέγει όμως το ψηφοδέλτιο ενός Ισλαμικού κόμματος, του Εναντά. Αυτό μήπως σημαίνει ότι η παρουσία της γυναίκας σε ένα κόμμα έρχεται σε αντίθεση με το Ισλάμ. Αντιθέτως, η απάντηση είναι όχι. Τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν να συμβιώσουν. Το Ισλάμ μπορεί να συνοδεύσει ε, τη γυναίκα στην πορεία της την πολιτική της πορεία ως πλήρες μέλος της πολιτικής ζωής. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, σας είμαι ευγνώμων για την τιμή που μας κάνετε σήμερα. Σας είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να παραστούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Είμαστε προσκεκλημένες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ε, για εμάς και είναι και μεγάλη τιμή που έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε το λόγο εδώ σε αυτό το βήμα. Είναι γεγονό ότι οι γυναίκε δεν κατέχουν πολλέ θέσει λήψη αποφάσεων στι χώρε μα. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη δική μου χώρα, την Τινησία, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μεταβατικό στάδιο, το οποίο έχουν γνωρίσει όλε οι χώρε τι οποίε έχουν σημειωθεί και έχουν ε, εκδηλωθεί επαναστάσει. Πρέπει να πούμε και να καταλογίσουμε στα θετικά της υπόθεσης ότι στη Ισία μετά τις εξελίξεις της Ραγδαίας δεν υπήρξε χάος. Αυτό το αποφύγαμε. Έχουμε λοιπόν το πολιτικό μας εγχείρημα. Έχουμε το κόμμα Ενάντα, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση σήμερα και στην ανοικοδόμηση της χώρας μας. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε ε, εκ των προτέρων. Δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στις κρίσεις μας. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε ε, πού θα καταλήξει ε, η κυβερνητική συμμαχία, ο κυβερνητικός συνασπισμός. Έχουν εκδηλωθεί ανησυχίες σύμφωνα με τις οποίες θα τερίσει ο στεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μου μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Εγώ διαφωνώ. Το έναν χαντά είναι ένα κόμμα το οποίο απαριθμεί πολλές γυναίκες στις τάξεις του και μία από αυτές τις γυναίκες, η υποφαινόμενη, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής για τους μάρτυρες και τους τραυματίες, για τη γενική αμνηστία. Είμαι και πρόεδρος και σε άλλη επιτροπή επίσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η θέση της γυναίκας σήμερα ενδυναμώνεται στην Τινησία, η παρουσία της ενδυναμώνεται στην Τινησία, παρόλο που οι γυναίκες στην κυβέρνηση είναι λίγες και δεν τους δόθηκαν υπουργικά χαρτοφυλάκια. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κίνημα. Έχουμε εξελίξεις πολλές ε, ο κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί ενδεχομένως να ε, αντιμετωπίζει εμπόδια, να πέφτει σε ενέδρες, να εκτροχιάζεται ενδεχομένως. Όλα αυτά οφείλονται στη μεταβατική περίοδο. Θα κάνει το πάνω όμως για να βελτιώσει την κατάσταση ώστε να έχουν καλύτερο μέλλον και οι άνδρες και οι γυναίκες στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, η επόμενη ομιλήτρια. Συνεχίστε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε. Θα ήθελα να μιλήσω γαλλικά για αλλαγή, παρόλο που είμαι εξαιρετικά περήφανη για την αραβική γλώσσα. Μου αρέσει όμως η εναλλαγή και η γλωσσική πολυμορφία και γι' αυτό προτιμώ μετά τα αραβικά να μιλήσω τώρα εγώ γαλλικά. Η Αραβική Άνοιξη πράγματι ήταν σημείο καμπής για όλες τις αραβικές χώρες σε όλα τα επίπεδα. Ο ρυθμός έλευσης των μεταρρυθμίσεων επιταχύνθηκε, αυξήθηκε. Δεν είχαμε ε, αστάθεια στο Μαρόκο, ε, χώρα από την οποία κατάγομαι, είχαμε περισσότερες διεκδικήσεις για περισσότερη διαφάνεια, για περισσότερη ε, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, από το 2002 μέχρι και σήμερα η γυναίκα είναι όλο και περισσότερο παρούσα με την Αραβική Άνοιξη εξετάστηκε και το νέο σύνταγμα το οποίο παρουσιάζει πρόοδο ως προς τις, ε, τα θέματα των γυναικών. Αλλά ήδη από το 2002 είχαν αρχίσει να δρομολογούνται όλα αυτά τα θέματα υπέρ των γυναικών. Το ποσοστό που πήραμε δεν είναι ε, τόσο μεγάλο, ωστόσο ε, είναι αρκετά ε, σημαντικό και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Έχουμε το άρθρο 19 του νέου συντάγματος, το οποίο επιμένει για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν εφαρμόζεται πλήρως, ωστόσο το νέο σύνταγμα μόλις πρόσφατα υιοθετήθηκε. εδώ και αρκετό καιρό, πολύ καιρό θα έλεγα, ακόμα και πριν από την ε, Αραβική Άνοιξη, οι γυναίκες στο Μαρόκο ε, καταλαμβάνουν διάφορα αξιώματα, έχουν καταλάβει διάφορα αξιώματα, έχουμε γυναίκες δημάρχους, διευθύντριες και μάλιστα ο πιο νέος δήμαρχος σε πόλη ε, στη χώρα μου είναι γυναίκα. Και μάλιστα ο, το πιο νέο μέλος του Κοινοβουλίου στη χώρα μου είναι γυναίκα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι, ε, αναδεικνύουν το δημοκρατικό εγχείρημα που έχει αναλάβει η χώρα μου. Ε, κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, διανύουμε όλη αυτή την απόσταση. Δεν την έχουμε καλύψει ακόμα. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε εδώ μετα... μαζί με εσά για να μοιραστούμε τις ιδέες μας, να εμπλουτιστούμε από τις δικές σας και αντιστρόφως. Σίγουρα, όπως είπαμε ε, και σήμερα το πρωί, μπορεί να υπάρχουν πολιτιστικά, ε, πολιτιστικοί περιορισμοί. Υπάρχει και ο περιορισμός των συνηθιών, διαφορετικές είναι οι συνήθειες. Δεν είμαστε εδώ για να αντιγράψουμε τυφλά τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Είμαστε εδώ για να βρεθεί μια συνένεση, για να υπάρξει μια ανταλλαγή ιδεών, ώστε να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας στον αραβικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα η θέση της γυναίκας στο Μαρόκο, ε, χώρα την οποία εγώ εκπροσωπώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Μπορείτε να μας πείτε και το όνομά σας, παρακαλώ. Η κυρία Σακέρ Σαϊντά, μέλος του Κοινοβουλίου στο Μαρόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρώτη πρόεδρος της κοινότητας. Ενώ η προηγούμενη ομιλήτρια λέει από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση της Τινησίας και πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Πολιτικές Ελευθερίες. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής σας. Παρακαλούμε η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Ναϊμά Μοχάμεντ Αλχάμι, μέλος του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου της Λιβύης. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κογκρέσου αυτή, αυτού και μέλος της Επιτροπής για τη Νεότητα, για τη Νεολαία και για τα Αθλήματα. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ε, καλησπέρα. Και να σας πω ότι στη Λιβύη η κατάσταση διαφέρει άρδιν συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Βορείου Αφρικής. Για δεκαετίες ολόκληρες στη Λιβύη ζήσαμε σύμφωνα με την εξής αρχή. Όσοι προσχωρούν σε κόμμα είναι προδότες. Σήμερα όμως ε, βιώνουμε την εμπειρία της πολυκομματικότητας και από το Φεβρουάριο την επανάσταση αυτή ε, η γυναίκα έχει αλλάξει ρόλο και έχει πραγματικά επαναστατήσει δίπλα-δίπλα με τον γιο της, τον σύζυγό της, ε, τον πατέρα της. Η γυναίκα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ε, αυτές τις εξελίξεις και σήμερα οι γυναίκες μπορούν να είναι βουλευτές, μέλη του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου, το οποίο είναι μια συντακτική συνέλευση και έχει ως καθήκον την κατάρτιση, σύνταξη του συντάγματος και ε, έχει και την υψηλή επιτροπή, ε, των, ε, ύπατη επιτροπή αν θέλετε, των εκλογών. Σήμερα λοιπόν η γυναίκα στη Λιβύη βλέπει τα δικαιώματά της να ε, υποστηρίζονται. Έχουμε γυναίκες προέδρους σε ορισμένες επιτροπές του Κογκρέσου, έχουμε ορισμένες γυναίκες υπουργούς, το χαρτοφυλάκιο το αντίστοιχο είναι, ε, έχει ανατεθεί σε γυναίκα, έχουμε γυναίκες δικαστές, Έχουμε λοιπόν ορισμένες γυναίκες σε ορισμένες θέσεις ε, στα διάφορα κέντρα εξουσίας στη χώρα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πρόοδος είναι μια καλή εξέλιξη για τις γυναίκες. Σήμερα λοιπόν ε, θα έλεγα, όπως γνωρίζετε, το 17% των μελών του Κογκρέσου, της Βουλής δηλαδή της Λιβύης, είναι γυναίκες. Και αυτό το ποσοστό δεν είναι κι άσχημο συγκριτικά με τις άλλες χώρες και αν λάβουμε και υπόψη μας την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας. Θα ήθελα να πω ότι ο γυναίκα είναι και ο πιο νέος βουλευτής ε, στη Βουλή μας. Το νεότερο μέλος λοιπόν της Βουλής μας είναι γυναίκα. Δύο αντιπρόεδροι επιτροπών είναι γυναίκες καθώς και η εισηγήτρια. Στο Γενικό Εθνικό Κογκρέσο που είναι η Βουλή μας εκπροσωπούνται πολλά και διαφορετικά κόμματα. Ορισμένες γυναίκες εξελέγησαν διότι είχαν εγγραφεί στο ψηφοδέλτιο των πολιτικών ε, κομμάτων. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του που τοποθετούνται τα πολιτικά κόμματα στο πολιτικό φάσμα, όλες αυτές οι γυναίκες από τα διάφορα ε, κόμματα έφτιαξαν, σύστησαν ένα μπλοκ γυναικών ώστε να προωθήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους μέσα στο Γενικό Εθνικό Κογκρέσο, μέσα στη Βουλή, ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην κατάρτιση, στη σύνταξη του συντάγματος. Εξού λοιπόν και η περηφάνεια που νιώθουμε. Είμαστε πολύ περήφανες που βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί απόδειξη όλων αυτών των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας ως προς την εκπροσώπηση των γυναικών στη δημόσια ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο αν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις μαρτυρίες σας, λέει η κυρία Κιλ Νίλσεν. Θα ήθελα να επανέλθω την κατάσταση στη Τινησία, γιατί ήμουν μέλος της αποστολής, της ανταπροσωπείας μας στη Τίνιδα πριν από αρκε... κάποιο καιρό. Ακούσαμε με προσοχή και με ενδιαφέρον ε, τις γυναίκες που είναι μέλη της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης και την Αντιπρόεδρο ε, από το κόμμα Έναν Χαντά, το ίδιο κόμμα ε, στο οποίο ανήκετε και εσείς, η πρώτη ομιλήτρια. Μιλήσατε πολύ για τη θρησκεία προηγουμένως στην παρέμβασή σας. Αναφέρομαι στην πρώτη ομιλήτρια βεβαίως. Και το θεωρώ το λογικό. Όποιο και αν είναι ε, το θρησκευτικό δόγμα στο οποίο προσχωρεί κανείς, ε, πάντοτε έχει γίνει θέμα συζήτησης και εξέτασης η θέση των γυναικών και στο χριστιανισμό και στον Ινδουισμό και ε, στον Ισλαμισμό μεταξύ άλλων. Πάντοτε η θέση της γυναίκας είναι κάτι το σημαντικό ε, στη σφαίρα της θρησκείας. Εγώ τίνω να πω ότι ε, καμία θρησκεία, σε καμία θρησκεία δεν αρέσουν πραγματικά οι γυναίκες, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, εν πάση περιπτώσει. Όταν λοιπόν συνάντησα τη συναδέλφου σας στην Εθνική Συντακτική Συνέλευση κατά την παραμονή μου στην Τίνητα πρόλεγου καιρού, ε, έμαθα για μια συζήτηση, για ένα διάλογο πολύ σημαντικό και σας ερωτώ ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις ως προς αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ε, ε, ε, εκκρεμούσε το ερώτημα το κατά πόσο το Σύνταγμα της Τινησίας θα αναφερθεί ρητός ότι επίσημη θρησκεία της ε, Τινησίας είναι η, ε, ε, το Ισλάμ. Αυτό ισχύει και αλλού στην Ευρώπη. Άλλωστε, επίσημη θρησκεία της περιφέρειάς μου εμένα στη Γαλλία είναι ο καθολικισμός. Εγώ είμαι από τη Βρετάνη και ο καθολικισμός είναι εξαιρετικά παρόν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ήταν το εξής. Στο Σύνταγμα θα γράφατε αν θα γράφατε ότι η επίσημη θρησκεία της ε, Τινησίας είναι το Ισλάμ ή αν θα γράφατε ότι το Ισλάμ είναι η πηγή από την οποία εκπορεύεται ο νόμος. Και η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο διατυπώσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για τα δικαιώματα τα ατομικά και πιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα των γυναικών. Ποιε είναι οι εξελίξεις λοιπόν ως προς αυτό το δίλημα, ε, προς τα που ε, κινείται η πλάστικα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο πήρε η κυρία Κιλνίλσεν που ήταν παρούσα, που συμμετείχε και αυτή στο ταξίδι μαζί με την κυρία Κώστα και εμένα. Η κυρία Κώστα έχει κάτι να προσθέσει. Φυσικά είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να ακούει κανείς απευθείας τις ε, βουλευτές να μιλούν εκείνες κάτι που είχε ήδη συμβεί στις συναντήσεις μας. Πρώτα απ' όλα η επίγνωση και η ένταση με την οποία ζουν αυτή την περίοδο στη χώρα τους οι γυναίκες, γνωρίζοντας ότι θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Συχνά ο ρόλος τους από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και της Ευρώπης παρουσιάζεται διαφορετικά. Δεν γίνεται αντιληπτό πόσο οι ίδιοι συνειδητοποιούν ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για να ενισχύσουν την θέση τους ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπε η βουλευτής από την Λιβύη ότι ακόμη και μεταξύ διαφορετικών κομμάτων υπάρχει μία ε, συνένωση των γυναικών, συνασπισμός τροποντινά με σκοπό να βελτιωθεί η μεταρρύθμιση του συντάγματο και η κοινοβουλευτική θέση των γυναικών μέσα από την νομοθεσία. Αυτό ώστε οριζόντια σε όλα τα κόμματα οι γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη εξουσία μέσα από το Σύνταγμα το οποίο να εγκριθεί. Ακόμα και στην Τινησία συζητήθηκε αυτό, παρόλο που ήταν κάπως πιο προβληματικό. Γι' αυτό και θα ρωτήσω τις γυναίκες από την Τινησία κατά πόσον και στη δική τους τη συντακτική συνέλευση <clears throat> μεταξύ γυναικών με διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες το συζητήσαμε και από την πλευρά της πλειοψηφία και της αντιπολίτευσης κατά πόσον λοιπόν υπάρχει προσπάθεια να διασφαλιστεί μια κοινή πρόταση για την ισότητα των γυναικών για τους νόμους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάστασή τους, ακόμη και πέραν των στενών κομματικών προτεραιοτήτων. Τώρα, για τα όσα αναμένουν από την Ευρώπη, ποιες είναι οι προσδοκίες τους, διότι εμείς έχουμε περικοπές τους πόρους και στις εταιρικές μας σχέσεις, και στις διμερείς με τις επιμέρους χώρες, με το Μαρόκο και την Τινησία αλλά και την Αίγυπτο, όπου τις μέρες αυτές από την ε, ομάδα μου λόγω χάρη υπάρχει επίσκεψη στην Αίγυπτο για τη στήριξη της όλης διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς θεωρείτε σημαντικότερες Είναι σωστή η διαδικασία αυτή που ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η αλληλεγγύη δική μας να έχει απόκριση την ε, απήχηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προστασία τους και στα κοινοβουλευτικά σώματα και στις κυβερνήσεις των χωρών σας. Σας ευχαριστώ πολύ και προτού να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε θα ήθελα να προσθέσω μια δική μου ερώτηση. στις χώρες σας ε, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, ε, επανάσταση, μεταρρύθμιση, πώς θέλει να το πει κανείς. Εσείς ε, οι γυναίκες αγωνιστήκατε εξίσου θαραλέα με τους άντρες για να αποκτήσετε την ελευθερία σας. Τώρα εκ των υστέρων δεν είναι εξίσου αυτονόητο ότι θα έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες, ότι θα έχετε ε, εξίσου καλή εκπροσώπηση κλπ. Είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά ήθελα να μου απαντήσετε πώς νιώθετε. Είσαστε απογοητευμένες εφόσον μαζί με τους άντρες αγωνιστήκατε για τη δημοκρατία και την ελευθερία και εκ των υστέρων βλέπετε ότι οι συνθήκες σας δεν είναι εξίσου καλές. Η δική μου πρόπτικη είναι λάθος. θα χαρώ πολύ αν μπορεί κάποια από εσά να μου απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Σας δίνω λοιπόν και πάλι το λόγο. Μπορείτε να μοιραστείτε το χρόνο όπως θέλετε. Παρακαλώ λοιπόν να απαντήσετε στις ερωτήσεις ε, που σας θέσαμε. Ευχαριστώ. Εγώ ως μόνο εκπρόσωπος της Τινησίας πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσω. Γι' αυτό που είπατε προηγουμένως, ε, θέλουμε να επιμείνουμε στο γεγονός ότι διατηρήσαμε το πρώτο άρθρο του προηγούμενης εκδοχής του συντάγματος. Σε καμία περίπτωση δεν θελήσαμε να πούμε ότι η Σαρία θα είναι η μόνη πηγή ε, νομοθετικής έμπνευσης στην Τινησία. Αυτό συζητήθηκε εκτός κοινοβουλευτικού σώματος. Στη συντακτική συνέλευση κάποιοι αντέτειναν ότι η Σαρία θα πρέπει να είναι η πρώτη ή η μόνη πηγή για την έμπνευση του συντάγματος. Το δικό μας κόμμα ουδέποτε όμως αποδεχτεί τέτοια αρχή. Όλοι συμφωνούμε ότι το πρώτο άρθρο ορίζει την Τινησία ως χώρα αραβική με επίσημη γλώσσα τα αραβικά και επίσημη θρησκεία το Ισλάμ. Το άρθρο αυτό δεν το αγγίξαμε. Αυτή η επιλογή είχε ήδη γίνει και έχει τύχει πλήρους συνένεσους. Νομίζω όταν μιλάμε για την Σαρία υπάρχει μια ενός φοβία, κάτι που όλους σας τρομάζει, αλλά ουδέποτε προτάθηκε κάτι τέτοιο στην Τινησία. Πώς λοιπόν να δούμε αυτή τη συζήτηση ως ελιγμό. Μια απλή συζήτηση ήταν και ανταλλαγή απόψεων. Όπως λόγου χάρη όταν τα κόμματα ε, στις εκλογές που θα κερδίσουν, εάν κερδίσουν τα Ισλαμιστικά κόμματα, εκεί θα αποδυναμωθεί η θέση της γυναίκας. Αλλά εδώ μιλάμε για προεκλογική εκστρατεία. Κάποιοι φοβούνταν την ε, νίκη των κομμάτων με θρησκευτικού ε, προσανατολισμού Φοβούνταν οποιαδήποτε στήριξη της ε, θρησκεία την, την Ισία. Το προηγούμενο καθεστώς είχε εγκαθιδρύσει αυτού του είδους το φόβο. Γι' αυτό και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα από κάποιους πολιτευόμενους της αντιπολίτευσης κατά την προεκλογική εκστρατεία. Εδώ λοιπόν υπάρχει σαφώς συνένεση ως προς τη θρησκεία. Διατηρήσαμε και διαφυλάξαμε αυτό που περιλαμβανόταν στο Σύνταγμα το 1959. Συνένεση ως προς την παρουσία της θρησκείας και βεβαίως ουδέτερος χαρακτήρας στους τόπους λατρείας. Δεν θα πρέπει να γίνουν ε, χώροι πολιτικής ή θρησκευτική προπαγάνδας. Αυτό εκφράζεται ρητός στο Σύνταγμά μας. Πέραν της ισότητας ανδρών και γυναικών, η ισότητα αυτή θα πρέπει να διαφυλάσσεται από το Σύνταγμα. Απέτηση όλων των ε, πολιτών. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να μην σεβαστεί αυτή την ισότητα. Ως γυναίκες βουλευτές από οποιοδήποτε κόμμα η πολιτική οικογένεια και αν προερχόμαστε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συμπαγές σώμα γυναικών στη Πουλή, ώστε να προασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών. Απλώς ενώσαμε τις δυνάμεις μας εντός Βουλής, διότι το Σύνταγμα προφανώς απαγορεύει την ε, προσχώρηση σε δύο διαφορετικά κόμματα ή δύο διαφορετικά, διαφορετικούς συνασπισμούς κομμάτων. Η αρχή που μας καθοδήγησε ήταν η αρχή συντονισμού των προσπαθειών μας, όποια και αν είναι η κομματική μας προέλευση. Τώρα τι προσδοκίες έχουμε από την Ευρώπη. Για μας στην Τινησία η Ευρώπη είναι ένας εταίρος. Έχουμε σχέσεις ε, εγκαθιδρυμένες, παραδοσιακές με την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να αντιγράψουμε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά έχετε προχωρήσει περισσότερο από εμά στην οδό της δημοκρατίας, του εκδημοκρατισμού και θέλουμε να προχωρήσουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο. Θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε τις δημοκρατικές αξίες, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τις οικουμενικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα για την κοινωνία της Τινησίας. Βάσει αυτών των δεδομένων πρέπει να ανταλλάξουμε μεταξύ μα γνώσει και εμπειρίε ώστε να υποφεληθούμε μένα από τι εμπειρίε των ΔΕ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Είναι μεγάλη μας χαρά να σας ε, απευθυνόμαστε στην αίθουσα αυτή. Η κατάσταση διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. Εμείς οι γυναίκες από το Μαρόκο δεν χρειάστηκε να κατέβουμε στους δρόμους όπως οι γυναίκες των άλλων χωρών. Ο βασιλιάς μας ε, διέταξε συνταγματική μεταρρύθμιση και εμείς κατεβήκαμε στους δρόμους για να στηρίξουμε αυτό το βασιλικό αίτημα ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα, η ισονομία και βάσει του άρθρου 19 του συντάγματος. Όταν συζητούμε για ισότητα και το συζητήσαμε και σε προηγούμενη συνεδρίαση, κάποιοι συνάδελφοι ίσως μας απαντήσουν ότι αποσπάσαμε 60 έδρες λόγω του συστήματος ποσοστώσεων. και 7 σε τοπικό επίπεδο. Μας λένε ότι ακόμα και στην Ευρώπη Υπάρχουν σχετικές εξελίξεις. Εγώ βλέπω νεαρές ε, βουλευτές στην αίθουσα και θα ήθελα να υποφεληθώ από τις δικές σας γνώσεις για την Ευρώπη, διότι οι γυναίκες στο Μαρόκο ε, κέρδισαν ένα σημαντικό αριθμό εδρών, όμως δυστυχώς η νοοτροπία των ε, ανδρών είναι αυτή που κυριαρχεί στο τοπίο. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να λάβουν το ρόλο του μπροστάρι στον δρόμο της δημοκρατίας. Είμαι η Μούχνα Φατιά, βουλευτής από το Μαρόκο και εισηγήτρια στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και Νομοθετικής Μεταρρύθμισης. Λέγομαι Σελίμα Μαφαραζή, είμαι βουλευτής της Αντιπολίτευσης Αυθεντικότητα και ε, Πρόοδος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συνταγματικών Δικαιωμάτων στο Μαρόκο. Να προσθέσω τα εξής τα προβλήματα που ε, έχει να αντιμετωπίσει η γυναίκα είναι η πατριαρχική κοινωνία και οι αλλαγέ ε, οι πολιτισμικέ. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία για να προστατευτούν οι γυναίκε στο σύστημα. Ποσοστώσεων, όπω είπατε, δεν πέτυχε στην Αίγυπτο με 2% των γυναικών να εκλέγονται σε μια χώρα σαν την Αίγυπτο. Δεν είναι δίκαιο αυτό για την ε, Αίγυπτο. 2% είναι πάρα πολύ λίγο. Ακόμη και για την Ευρώπη και τι ΗΠΑ είναι χαμηλά τα ποσοστά. Το πρόβλημα λοιπόν που τίθεται είναι η πατριαρχική κοινωνία. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Να ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση. Διότι το σύστημα ποσοστώσεων στο Μαρόκο πέρασε από δύο βουλευτέ, ε, γιατί βρισκόμαστε στη δεύτερη θητεία πλέον, σε τέσσερι, 30 και τώρα έχουμε φτάσει στι 60. 60 γυναίκε ε, στι εκλογικού καταλόγου. Επτά γυναίκες ε, κατάφεραν να εκλεγούν. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα πραγματικό πρόβλημα. Βεβαίως στο Μαρόκο. Το θέμα είναι ο ρόλος των οικογενειών. Ε, το οικογενειακό δίκαιο δηλαδή Τώρα μπορεί μια γυναίκα να ζητήσει διαζύγιο χωρίς ε, να επικαλέσει συγκεκριμένα αίτια. Προηγουμένως ε, έπρεπε να υπάρχουν σοβαρά αίτια, όπως η εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, ε, η εγκατάλειψη από το σύζυγο και το καθεξής. Εδώ μπορεί να πει απλώ θέλω να χωρίσω γιατί δεν μου αρέσει ο σύζυγό μου. Μπορεί να αλλάξει η χώρα κατοικία, μπορεί να αλλάξει δουλειά. Βεβαίω έχουμε μόνο μία γυναίκα υπουργό Ω κόμμα αντιπολίτευση δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Ελπίζουμε όμω ότι οι γυναίκε θα πολεμήσουν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανδρών από τα μέσα μαζική επικοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει με τι γυναίκε, ακόμη και όταν είναι φορεί τη κοινωνία των πολιτών. Όλε οι προσπάθειε που καταβάλουν οι γυναίκε δεν σημαίνει ότι προβάλλονται από τα μέσα. οι προσπάθειε που γίνονται από του άντρε μπορεί να είναι λιγότερε, αλλά προβάλλονται το πολλαπλάσια. Έτσι λοιπόν οι γυναίκε θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν πολλή δουλειά μπροστά του για να καταφέρουν να πείσουν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι και η καταπολέμηση των γυναικών τη ίδια τη γυναίκε. Καμιά φορά οι γυναίκε υποβάλλουν υποψηφιότητα και οι υπόλοιπε γυναίκε δεν τι ψηφίζουν. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι υπάρχει, πρόβλημα δημοσκοπήσεων, πρόβλημα Βεβαίω η ψηφοφορία μυστική. Όμω, όταν θέτουμε το ερώτημα στου πολίτε, διότι στη Βουλή ρόλο των βουλευτών δεν είναι μόνο η νομοθεσία, η διακυβέρνηση, η παράλληλη διπλωματία, αλλά και η συνομιλία επαφή με τους πολίτες. Οι βουλευτές λοιπόν μέσα από τις επαφές τους με τους πολίτες καταφέρνουν να δουν τι ανεπάρκειε του συστήματο και τι ανάγκε των μακητών Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες δεν εμπιστεύονται απολύτω τι άλλες γυναίκες. Αυτό δεν αφορά μόνο το Μαγκρέπ, τη Βόρεια Αφρική. Αυτό ε, μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως ε, τους ε, συλλόγους, τους επαγγελματικούς συλλόγους. στην Καζαμπλάνκα, λόγω χάρη, έχουμε μόνο 800 γυναίκες. Πρέπει λοιπόν οι γυναίκες να ευαισθητοποιηθούν. Τα ισχυρά κόμματα πρέπει να δουν αν μπορούν να βάλουν σε ενό εκλογικού καταλόγου μια γυναίκα. Το σύστημα ποσοστώσεων κάθε, κάποιες φορές υποβαθμίζει το όλων των γυναικών. Γιατί δεν πείθεται όμω και η κοινωνία των πολιτών, γιατί δεν πείθονται οι υπόλοιπε γυναίκε. Κάπω έτσι έχουν τα προβλήματα και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε, να αγωνιστούμε και να πείσουμε. Ευχαριστώ. Is it else? Σας ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Με λένε Σελιμά Φαραζή και είμαι μέλος της Βουλής, λέει η προηγούμενη ομιλήτρια. Εμένα με λένε Χαλενόρφη και είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα υγείας και μέλος της Επιτροπής για τους παλέμαχους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εκπροσωπούμε τις γυναίκες της Λιβύης δεν έχουμε απογοητευτεί με το αποτέλεσμα αυτό. Αντιθέτως, είναι μεγάλη χαρά για μας, μεγάλη ευχαρίστηση. Πρόκειται για το πρώτο συντακτικό κογκρέσιο το οποίο εξελέγει στη Λιβύη για πρώτη φορά στα χρονικά της. Ακούσαμε ότι το ποσοστό των γυναικών στην Ευρώπη ανέρχεται στο 5% στην αρχή και έχει φτάσει τώρα στο 35% μετά από τόσα πολλά χρόνια εκλογών, επαναλαμβανόμενων εκλογών. Ενώ εμείς στη Λιβύη με την πρώτη εκλογή φτάσαμε στο 17%. Δεν είναι και λίγο. Νομίζω ότι ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε ότι η γυναίκα θυσίασε πολλά κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και δεν κατάφερε να επιτύχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι οι άνδρες θυσίασαν πολλά. Έγιναν μάρτυρες. Η Λιβύη είναι χώρα 50.000 μαρτύρων, θυμάτων και η πλειονότητα ήταν άνδρες. Σε αυτή τη μάχη για το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών. Θέλουμε αυτά να κατοχυρωθούν συνταγματικά. επιθυμούμε τα επόμενα χρόνια πράγματι να καταλήξουμε σε ισότητα, αν όχι πλήρη τουλάχιστον στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μεταξύ ανδρών και γυναικών και ισότιμη εκπροσώπηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτού να κλείσουμε, θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπα. Που είπατε ότι ε, παλεύετε εσείς, ε, αγωνίζεστε στις ε, χώρες σας για την δημοκρατία και την ελευθερία. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο αγωνιζόμαστε για την ισότητα. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε 34% γυναίκες βουλευτές. Είναι αρκετά καλό ποσοστό αυτό, διότι ο μέσος όρος των κρατών μελών είναι 22%. Ε, σε κάποιες χώρε το ποσοστό είναι χαμηλότερο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν απομένουν πολλά να γίνουν, πρέπει να γίνουν πολλά, όπως άλλωστε σε όλο τον κόσμο. Γιατί λοιπόν ε, έχει έτσι η κατάσταση, επειδή ζούμε σε πατριαρχικές δομές. Οι άντρες λοιπόν έχουν αρκετή εξουσία, οι άντρες εκλέγουν τους έντρε. οι άντρες διορίζουν άντρες και αυτή η δομή υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να διατηρήσουμε τη δομή αυτή, θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό, είτε βρισκόμαστε στην Αφρική είτε στην Ευρώπη. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που μπορέσατε να έρθετε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αφιερώσατε το χρόνο σας. Ε, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι την εβδομάδα που θα παραμείνετε εδώ να ε, μπορέσετε να μάθετε από τις δικές μας εργασίες και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και ε, με τα λόγια αυτά κλείνει η σημερινή μα συνεδρίαση. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί στι 9.